Mes chers collègues, bonjour. Καλημέρα συνάδελφοι. Σας εύχομαι σε όλους καλή αρχή σχολικής χρονιάς με ισχυρές δεσμεύσεις. Μία από τις πρώτες δεσμεύσεις που θα πρέπει να αναλάβουμε είναι να απαγορευτούν τα πλαστικά μπουκάλια. Κοιτάξτε κύριε Ρικέ, δίνω το παράδειγμα. Έχω γυάλινο μπουκάλι. Ευχαριστώ και όλους τους διερμηνείς που είναι εδώ μαζί μας. Ελπίζω οι διακοπές σας να ήταν καλές και ελπίζω να έχετε έρθει δρυμύτεροι. Βικτόρ, μιλάω υπό την δική σου εποπτεία. Θα περάσουμε σήμερα μια πολύ δύσκολη χρονιά. Οι δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουμε θα είναι φιλόδοξες και την ίδια ώρα θα πρέπει να επιτύχουμε τα αποτελέσματα. Σκοπός μας είναι να αλλάξουμε τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Σκοπός μας είναι οι μεταφορές να μην είναι μία ταλαιπωρία, αλλά να είναι μεταφορές αρμονικές, οι οποίες θα επιλέγονται από τους πολίτες μας και δεν θα τις ε, ε, υποστούν χωρίς να έχουν απολύτως καμία επιλογή. Ξεκινάω με την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχει καμία παρατήρηση, υιοθετείτε. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Είστε τυχεροί σήμερα. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις της Προέδρου. Όσον αφορά τώρα τα πρακτικά, νομίζω ότι μπορούμε να τα υιοθετήσουμε, εκτός αν υπάρχουν αντιρρήσεις. Πρόκειται για τα πρακτικά της 10 ε, Ιουλίου και της 24 η Ιουλίου. Και έχουμε ήδη φτάσει στο σημείο 4, Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, όλα τα τμήματα, αγαπητοί συνάδελφοι. Το σημείο αυτό το είχαμε ήδη προσεγγίσει πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο περίφημος προϋπολογισμός για το 2020. Κατόπιν θα συζητήσουμε και για τη γνωμοδότηση της δικής μας Επιτροπής που θα συζητηθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον εισηγητή και κατόπιν βεβαίως οι σκιώδεις εισηγητές θα πάρουν το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τοποθετηθεί. Υπενθυμίζω ότι θα ψηφίσουμε πολύ σύντομα τις τροπολογίες, δηλαδή Είχαμε δώσει μια ημερομηνία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, 9 Σεπτεμβρίου στις 3 είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Σύντομη προθεσμία, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τηρήσουμε το φιλόδοξο στόχο μας. Ο κύριος Ντάνιελ Φρόιντ. Καλημέρα σας, κύριε Σιγητά. Σας δίνω το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι για τις τροπολογίες που έχετε υποβάλει. Πολλές μπορώ να τις στηρίξω. Έχουμε σήμερα την δυνατότητα να έχουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων επ' αυτής της γνωμοδότησης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι χρειαζόμαστε μια πλήρη επισκόπηση για το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι ευρωπαϊκές μεταχώρες. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντικές ε, προκλήσεις που αφορούν το κλίμα, αφορούν την τήρηση των στόχων μας και των δεσμεύσεών μας υπό το φως της ε, Συνθήκης των Παρισιών. Πιστεύω πραγματικά ότι οι στόχοι και οι προκλήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναρχίσει η επεξεργασία του προϋπολογισμού αυτού, έχοντας κατά νου όλους αυτούς τους στόχους. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, αδυναμίες, οι προτάσεις ε, του Συμβουλίου είναι περικοπές, περικοπές ε, σε όλα τα τμήματα και για τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών μεταφορών που είναι όπως ξέρουμε όλοι ένας ε, βιώσιμος ε, τρόπος, ο πιο βιώσιμος τρόπος μεταφορών. Εγώ σαν εισηγητής ε, πρότεινα να επανέλθουμε για όλες αυτές τις περικοπές σε σημεία κλειδιά και όχι μόνο για τις υποδομές των ε, εμπορικών μεταφορών, αλλά και για τις ε, επιβατικές μεταφορές, ε, στηρίζοντας την βιώσιμη κινητικότητα και λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παραμέτρους που έχουμε δεσμευτεί να τηρήσουμε. Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και την στήριξη της χρηματοδότησης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης και την κλιματική διάσταση, το θέμα των επενδύσεων στην Ευρώπη. Οι στόχοι, επαναλαμβάνω, για το κλίμα πρέπει σε όλα τα σχέδια και προγράμματα επενδύσεων να λαμβάνονται υπόψη, καθώς και το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας. Αυτά είναι για μένα το, ε, τα γενικότερα περιγράμματα αυτού που θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Δεν έχουν συμπεριληφθεί οι διάφορες προτάσεις ε, του Ταμείου Συνοχής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υποβληθούν και κάποιες τροπολογίες που να λαμβάνουν υπόψη και αυτή τη συνιστόσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φρόντ. Ο κύριος Μαρινέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν και τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης που συνέταξε. Θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν να βασίσει την τελική της πρόταση για τον προπολογισμό του 2020 σε μια αξιολόγηση που θα αφορά το SEF, το Connecting Europe Facility, και τη δυνατότητα να δαπανηθούν τα χρήματα που έχουν ενταχθεί σε αυτό. Πώς όλες οι γραμμές, δηλαδή με άλλα λόγια, του ΣΕΦ, ιδίω τα χρηματοδοτικά μέσα, πώς η Κομισιόν ε, προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Γιατί το σημαντικότερο είναι να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί και όχι απλώ να καταλήξουμε στο τέλο τη διαδικασία, να, να συμπεράνουμε ότι κάποια κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να απορροφήσουν τα κονδύλια, να, να δαπανίσουν τα χρήματα που προβλέπονταν κτλ. κτλ. Δεν είναι αυτό ο στόχο. Τέλο, στο τέλο τη διαδικασία αυτή, όταν δηλαδή η Κομισιόν υποβάλλει την τελική τη πρόταση, να... Ε, υπάρχει μια αξιολόγηση για κάθε γραμμή και ποιε είναι οι δυνατότητε αξιοποίηση όλων των χρημάτων που είχαν δεσμευτεί ε, υπέρ του ΣΕΦ. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Με μια πραγματική αξιολόγηση της Επιτροπής έχετε δίκιο. Αυτό είναι ε, κάτι το πολύ σημαντικό. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών έχετε το λόγο. Εγώ... Αντικαθιστώ την κυρία Γκραπίνη ε, και θα σας διαβάσω αυτό που μου έδωσε στα ε, ρουμανικά. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να σας ζητήσω συγγνώμη που δεν παρευρίσκομαι στη σημερινή συζήτηση όσον αφορά το σχέδιο Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020. Θέμα για το οποίο εγώ είμαι σκιώδης συγγήτρια εκ μέρους των σοσιαλιστών, διότι συμμετέχω στην αποστολή στη Μολδαβία. Ανέλαβα το φάκελο αυτό από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, από την κυρία Ανταμόντα, που δεν είναι πλέον Ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την ε, εμπιστοσύνη που μου δείξατε αναθέτοντα μου το θέμα αυτό και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα για τον προπολογισμό του 2020. Οι μεταφορέ είναι πολύ σημαντικέ όταν μιλούμε για τον Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτο 2020, διότι εκεί προβλέπονται οι τρόποι με του οποίου θα λειτουργήσει η εσωτερική αγορά και προβλέπονται και οι τρόποι με τους οποίους θα μετακινούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Είναι θετικό το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2020 είναι υψηλότερος από εκείνο του 2019. Δυστυχώς όμως βλέπουμε το Συμβούλιο να προσπαθεί να περικόψει τα κονδύλια που δεσμεύονται και κατευθύνονται σε συγκεκριμένου τομεί του συστήματος ε, μεταφορών. Θεωρώ ότι πρέπει τα κονδύλια να αυξηθούν για τις μεταφορές, ώστε έως το 2050 να έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μηδενικές εκπομπές από τον κλάδο των μεταφορών προκειμένου να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που απορρέουν από την διάσκεψη των Παρισίων. Το σχέδιο αυτό δίνει περισσότερη έμφαση στην ποιότητα των έργων, όχι μόνο στην ποσότητα ή τις διαστάσεις. Όταν παρέχεται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επίσης, ε, προστίθεται πλέον ε, μια απέτηση για το κλίμα. Πιστεύω ότι στην Ευρώπη χρειαζόμαστε καλύτερη χρηματοδότηση για τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών, αλλά και για εκείνα τα έργα που προορίζονται για ε, την ε, επανέναρξη διασυνοριακών, διαπεριφερειακών, σειροδρομικών συνδέσεων που θα δώσουν καλύτερη συνδεσιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στη χρηματοδότηση των μέτρων που ε, ε, εξασφαλίζουν και βελτιώνουν την ασφάλεια των επιβατών και πρέπει επίσης να δώσουμε έμφαση στους ευάλωτους χρήστες όπως είναι οι πεζοί, οι ποδηλάτες κτλ. Το σχέδιο αυτό προσπαθεί να δώσει περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τους ε, δημόσιους διαγωνισμούς και τις προμήθειες στον τομέα των υποδομένων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό οι εργολάβοι να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και να παρέχουν ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια σε κάθε περίπτωση που ε, διανεργούνται τέτοιοι διαγωνισμοί. Έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες μαζί με συναδέλφους μου και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ε, αναμορφώσουμε στη σωστή κατεύθυνση τις προτάσεις της ε, Κομισιόν. Αύριο είναι η ψηφοφορία. Ε, η υποβολή για τις τροπολογίες είναι η 9η Σεπτεμβρίου. Σας καλώ και εγώ όλους έχετε να υποβάλλετε τις τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Τερές. Θέλω απλώς να σας πενθυμίσω κάτι που είναι σημαντικό. Ο προϋπολογισμός για τις μεταφορές προς το παρόν παραμένει. Και εδώ δεν αναφέρομαι στην πολιτική συνοχή ή την ΚΑΠ, για, την οποία, για τις οποίες δεν συμβαίνει το ίδιο. Προς το παρόν λοιπόν διατηρείται ως έχει. Θα δούμε τι θα γίνει με το Brexit. Και κοιτώ προς τον Ντομινίκ Ρικέ, ειδικό για τα θέματα αυτά. Μην ξεχνάτε όμως ότι ο προϋπολογισμός των μεταφορών δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση, είναι μία win-win κατάσταση για όλους. Κερδίζουμε για το κλίμα, κερδίζουμε στον τομέα των υποδομών. Όταν λοιπόν μειώνεται ο προϋπολογισμός των μεταφορών, θα πρέπει εμείς να πολεμήσουμε μέχρι να τον επαναφέρουμε διότι δεν είναι δυνατόν να υποχωρήσουμε και δεν είναι δυνατόν όπως προηγούμενες χρονιές να υπάρχουν περικοπές σε σχέδια και προγράμματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα και να έχουμε περικοπές της τάξης του 10%. Η μάχη μας λοιπόν παραμένει η ίδια, να παραμείνει ο προϋπολογισμός ως έχει, αλλά να τον κατευθύνουμε σε πιο σαφείς τομείς. Κύριε Ραμόν Βοζάντιας, τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι να επιμείνω στο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2020 πρέπει να είναι φιλόδοξος για τον τομέα των μεταφορών ως ε, ουσιαστικό ε, στοιχείο για την ελεύθερη κυκλοφορία και ατόμων αλλά και εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ο προπολογισμό πρέπει να λάβει υπόψη του τι πολιτικέ προτεραιότητε σε θέματα μεταφορών βεβαίω, οι οποίε κατά την άποψή μα είναι τρει. Καταρχά, να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Δεύτερον, να έχουμε μεγαλύτερε και καλύτερε επενδύσει και στην έρευνα και στην καινοτομία και να αυξήσει η ανάπτυξη τη κοινωνική συνοχή και τη εδαφική συνοχή για να μπορέσουμε να συνδέσουμε όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Ε, ένα από τα ουσιαστικά σημεία είναι ότι η χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε υποδομέ μεταφορών είναι ότι θα πρέπει ω βασικό στόχο να έχουν την αποτελεσματικότητα και να ε, εδραιώσουμε και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει σε θέματα κλίματο. Ε, πρέπει να υπάρχει αύξηση λοιπόν στη χρηματοδότηση γιατί είναι προσανατολισμένο σε αποτελέσματα και κυρίω στην αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων ε, στα οποία συμβάλλουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε. Θα ήθελα να σταθώ και σε κάποια ουσιαστικά σημεία το είπα και στη συζήτηση για τον προπολογισμό τον Ιούλιο, θα ήθελα να σταθώ στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος ε, συνδέεται απολύτως με τις μεταφορές πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση για τον τουρισμό και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη πρικοδότηση στον προπολογισμό ξεχωριστή για τον τουρισμό. Ε, ο τομέας του τουρισμού ε, δημιουργεί πολύ μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο, δημιουργεί ανάπτυξη, ε, σχέδια, θέσεις εργασίας και θεωρείται ως κάτι το οποίο ε, ε, έχει βοηθήσει και χώρες ε, σε περίοδο κρίσης. Ο τουρισμός μπόρεσε να βοηθήσει ώστε η κρίση να είναι λιγότερο έντονη ή και να βοηθήσει να υπερβούμε την κρίση. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και συγκεκριμένη μνήμα στο μηχανισμό Connecting Europe, που είναι ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο ζωτική σημασία για τον τομέα των μεταφορών και κυρίως για τους διαδρόμους του Ατλαντικού, της Μεσογείου κλπ. Ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να συνδέσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ε, εξασφαλίζοντας την ελευθερία και την οικονομική ανάπτυξή τους. Και ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε με μία ακόμα από τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει όχι μόνο εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών ε, την ε, μειωμένη χρήση άνθρακα και την ε, ψηφιοποίηση. Είναι και αυτές τεράστιες προκλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα που πρέπει να θεωρούνται και αυτές προτεραιότητα. Γι' αυτό ακριβώς και θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση για τα έργα και για τα συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία βοηθούν ε, τα θέματα της διακοπής της χρήσης άνθρακα και της ψηφιοποίησης. Αυτά νομίζω και από πολιτική σκοπιά θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά, έχετε δίκιο, διότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά τον τουρισμό. Ρομπέρ, καλημέρα. Ναι, χαίρομαι που σας βλέπω όλους μετά τις διακοπές. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ πιο πολύ στην γνωμοδότηση. Πρώτον, ο προεπολογισμός αυτός θα πρέπει να έχει μια προσέγγιση για τις άμεσες επενδύσεις και την προστιθέμενη αξία αυτών. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας για επενδύσεις και για δημιουργία νέων θέσεων αποσχόλησης. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να στηρίξουμε τον τομέα των μεταφορών και να στηρίξουμε κυρίως την ε, προστιθέμενη αξία του τομέα αυτού όσον αφορά αυτές τις βιώσιμες επενδύσεις. Invest EU, καθώς και τα προγράμματα που χρηματοδοτούν τις υποδομές αυτές στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να αναφερθούν. Είναι ουσιαστικό ένας βιώσιμος προϋπολογισμός ο οποίος πραγματικά θα στηρίξει την αξιοπιστία αυτών των προγραμμάτων που ήδη έχουν ξεκινήσει ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα στηρίξει τις επενδύσεις αυτές που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία αυτών των προγραμμάτων. Είδατε, πιστεύω, τις τροπολογίες μας, θα υποβάλουμε και άλλες όσον αφορά την στήριξη αυτών των επενδύσεων, της οικονομικής πτυχής αλλά και της βιωσιμότητας αυτών των προγραμμάτων. Θέλουμε αυτή η ισορροπία πραγματικά να τηρηθεί εδώ στην ε, Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ, Ρομπέρ. Εκ μέρους της ε, ΓΚΟΕ, η κυρία Κουτουρά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Φρόιντ, ο οποίος αναδεικνύει το μεγάλο ζήτημα της ανεπαρκούς χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών για όλα αυτά τα οποία, όλους τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Ε, εν όψη, μάλιστα ε, των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρέπει να εναρμονίζονται με τις διεθνείς μας δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Σε αυτή την μετάβαση του τομέα των μεταφορών θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να αποφύγουμε ορισμένες σημαντικές ανεπιθύμητες συνέπειες συγκεκριμένα. Οι πολιτικές που θα μας οδηγήσουν στη νέα πραγματικότητα θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη και την ανάγκη για προστασία των αδύναμων κοινωνικών ομάδων αλλά και τις ιδιαιτερότητες και σημεία εκκίνησης των κρατών και περιφερειών χωρίς βέβαια να είμαστε ελαστικοί στην επίτευξη των κλιματικών μας στόχων, αλλά θα πρέπει να υπολογίζεται και το κοινωνικό κόστος για να σχεδιάζονται παράλληλα τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα. Και αυτό είναι ζήτημα θεμελιώδου σημασία, γιατί αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή, χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων αλλά και περιφερειών. Διαφορετικά φοβάμαι ότι θα έχουμε αντιδράσει, οι οποίε μπορεί τελικά να υπονομεύσουν ε, ουσιαστικά τους στόχους μας. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό μας και στις μεταφορές και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στον τουρισμό ο οποίος λείπει από το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αλλά και από τη γνωμοδότηση που βρίσκεται σήμερα υπό συζήτηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το αίτημά μας διότι η σημασία του τουρισμού είναι τεράστια και για τις μεταφορές και φυσικά για την κοινωνική συνοχή αλλά πάνω απ' όλα για την ανάπτυξη και την ε, οικονομία. Διότι, για παράδειγμα, στα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, ο τουρισμός, ο οποίος είναι μια καθαρά εξωστρεφής δραστηριότητα, ήταν ο κεντρικός πυλώνας που στήριξε την οικονομία, οδήγησε την πατρίδα μας στην ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική, ενίσχυσε τις τοπικές κοινωνίες, ε, δημιούργησε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και φυσικά ενίσχυσε σημαντικά την εικόνα της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε για άλλη μία φορά να συμπεριληφθεί ο τουρισμός στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και φυσικά έχουμε συζητήσει και στην Επιτροπή μας για μια συνολική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Merci Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσω αμέσως το λόγο. Α, δεν θέλετε να πάρετε το λόγο. Κάποιος άλλος. Όχι. Τότε δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Μοντανιόν, να απαντήσει στις ερωτήσεις, κυρίως τις ερωτήσεις του εισηγητή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παραμείνει στον προϋπολογισμό που υιοθετήθηκε τον Μάιο. Το έχω πει, επανέρχομαι στο παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε ένα backloading των πληρωμών, πρόκειται για προγράμματα και σχέδια που έχουν πολύ λιγότερη ανάγκη χρηματοδότηση στην πρώτη τους φάση, στην αρχική φάση και πολύ περισσότερο στις μεταγενέστερες, στις πιο ε, οψιμές φάσεις. Πρόκειται επίσης για έναν προϋπολογισμό ο οποίος ε, δεν θα υποστεί περικοπές. Στηρίζουμε τις ε, προτάσεις σας να παραμείνουμε στον προϋπολογισμό εκείνων σε σχέση με τις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο που ανέρχονται στα 180 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνούμε λοιπόν με τις προτάσεις και θα τις στηρίξουμε. Όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και την προετοιμασία, τις δράσεις προετοιμασίας, γιατί υπήρξαν και κάποιες τροπολογίες που αφορούν αυτές τις δράσεις προετοιμασίας και τα πιλωτικά προγράμματα, ο δεύτερος γύρος δεν έχει ολοκληρωθεί φαντάζομαι όσον αφορά τις τροπολογίες. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν νέες τροπολογίες για τις νέες προτάσεις του Κοινοβουλίου. Θα εξετάσουμε όλες αυτές τις προτάσεις και τις τροπολογίες όταν ε, υποβληθούν στο σύνολό τους. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του κυρίου Μαρινέσκου και τις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, όλες οι εκκλήσεις μας που αφορούν το SEF, Connecting Europe Facility, αφορούν προγράμματα που είναι ήδη εν εξελίξη. Αν υπάρξει αύξηση και επιβεβαιωθεί για τις γραμμές προπολογισμού του ΣΕΦ, εμείς θα το στηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μοντανιό. Θέλω εδώ να πω ότι όσον αφορά τα θέματα τα δημοσιονομικά, η Επιτροπή προτείνει και εμείς αποφασίζουμε. Όταν μας λέτε ότι δεν θα αλλάξουμε τον προϋπολογισμό που είχαμε αρχικά προβλέψει, ε, λίγο με ενοχλεί αυτή, αν θέλετε, η θέση σας. Εσείς, όσον αφορά το, τους καλοκαιρινούς μήνες, τον καύσωνα, την εξάλληψη μεγάλου τμήματος της βιοπικιλότητας, φαίνεται να μην ταράζεστε πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι ο προϋπολογισμός αυτός, όσον αφορά τους πιο φιλόδοξους στόχους, αυτούς που αφορούν την COP21, αφορούσε των 9% των συνολικών κονδυλίων. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εμείς εδώ δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Η νέα επιτροπή, η πρόεδρος της νέας επιτροπής μίλησε για τη μειωμένη χρήση του άνθρακα, μίλησε για τις νέες προτεραιότητες και εμείς εδώ θα δώσουμε το ρυθμό που θέλουμε να ακολουθηθεί. Πραγματικά λοιπόν αυτά τα πιλωτικά προγράμματα θα πρέπει να στηριχθούν και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ο Ντάνιελ Φρέντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ συναδελφοί για τα σχόλια αυτά. υπομονώ και εγώ να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας για τις τροπολογίες και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε και την υπόλοιπη διαδικασία. Ευχαριστώ. Je Υπενθυμίζω ότι αύριο ψηφίζουμε. Να έχετε λοιπόν όλοι μαζί τις κάρτες σας, τις κάρτες ψηφοφορίας. Αύριο θα ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες που αφορούν τον προϋπολογισμό. Αύριο. Ψηφοφορία, λοιπόν. Και κατόπιν η υποβολή για την 9η Σεπτεμβρίου όσον αφορά την γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Σημειώσατε αυτές τις ημερομηνίε. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Θα περιμένουμε την ε, ψηφοφορία αύριο. Προχωρούμε στο σημείο 5. Ανταλλαγή απόψεων με τους συντονιστές ε, των διευρωπαϊκών δικτύων και μεταφορών. Είναι εδώ όλοι οι συντονιστές. Ελάτε να καθίστε εδώ δίπλα μου. Ο Κάρλος Σέση, ο οποίος είναι συντονιστής για τον διάδρομο του Ατλαντικού, ο κύριος Ματιό Γκρός, συντονιστής για το διάδρομο Ανατολική Μεσόγειος, Ανατολή Ανατολική Μεσόγειος και ο Πίτερ Μπάλας, ο οποίος είναι συντονιστής για τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Ο κύριος Έραλτ Ρόιτερς, ο οποίος είναι ο διευθυντής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στην DG Move. Καλώς ορίσατε.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 με την ακρόασή μας και την ανταλλαγή απόψεων. Συνεχίζουμε δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των διευρωπαϊκών δικτύων για τις μεταφορές, την αρχή της νέας μας θητείας. Μιλήσαμε για την πολιτική κινητικότητας και τον προϋπολογισμό μετά το 2020. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εξετάσουμε από κοινού και πολύ προσεκτικά αυτούς τους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου, τον άξονα κλειδί των διευρωπαϊκών δικτύων για τις μεταφορές. Θα ήθελα να ακούσουμε λοιπόν τους συντονιστές μας. Υπάρχουν εννέα διάδρομοι για όσους το έχουν ξεχάσει και έχουμε και τις οριζόντιες προοπτικές οι οποίες είναι στην καρδιά της νέας μας πολιτικής οι οποίες υιοθετήθηκαν το 2013. Δεν είμαι υπεύθυνη δεν ήμουνα μέλος του Κοινοβουλίου τότε, έχουν υλοποιηθεί από το 2013 μέχρι σήμερα. Πριν περάσουμε στο συγκεκριμένο θέμα των διαδρόμων, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βεβαίως θα τοποθετηθεί όσον αφορά την πρόεδρο υλοποίηση αυτών των ε, διευρωπαϊκών δικτύων, τις προοπτικές ε, για το μέλλον. Σας καλωσορίζω όλους λοιπόν και θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον Χέραλτ Ρόιτερς, ο οποίος θα μας κάνει μια πρώτη επισκόπηση για τις προκλήσεις. Κύριε Ρόιτερ, έχετε 12 λεπτά, ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στους συντονιστές, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν ο καθένας τον τομέα του, τις δυσκολίες και θα πρέπει πραγματικά σήμερα να μας μιλήσετε με μεγάλη ειλικρίνεια για τις δυσκολίες. Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Πολλές φορές υπάρχουν και διπλωματικές δυσκολίες. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε, να σας βοηθήσουμε. Μη φοβάστε, μιλήστε ελεύθερα. Θέλουμε όλοι να προχωρήσουμε και να υπάρξει πρόοδος. Κύριε Ρόιτερς, έχετε το λόγο για 12 λεπτά και βάζω και το χρονόμετρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη. Ε, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο σήμερα στην αρχή της νέας σας στη διάρκεια της οποίας θα μπορέσουμε να ε, συζητήσουμε αυτές τις πολιτικές, οι οποίες είναι πολιτικές υποδομών, αλλά και πολιτικές ε, προτύπων, επομένως και για την πολιτική μεταφορών εν γέννη. Θα δούμε λοιπόν και τις ε, διαπραγματεύσεις ε, για την αναθεώρηση, η οποία θα αλλάξει λίγο και θα συζητηθεί στην Επιτροπή σας ε, το 2021-2023, ελπίζω. Θα κάνω την παρουσίαση στα αγγλικά τώρα. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε γιατί ε, έχω προετοιμάσει τις ε, διαφάνειες στα αγγλικά. Όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι σε αυτή την πρώτη διαφάνεια έχουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα με όλες αυτές τις γραμμές με πράσινο, κόκκινο και μπλε τα οποία αντιπροσωπεύουν ε, τις εσωτερικές πλωτές οδούς, ε, αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους, ε, λιμένες, αεροδρόμια και όλα μαζί αποτελούν το διευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών. Και βεβαίως Αυτό περιλαμβάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ε, αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρόμων και σημεία σύνδεσης μεταξύ ε, των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης. Έχουμε ένα βασικό δίκτυο το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και ένα συμπληρωματικό δίκτυο το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ε, συνολικά μέχρι το 2050. Οι εκτιμήσεις για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών δείχνουν ότι θα δημιουργήσει πάνω από 1,6 επιπλέον ΑΕΠ και θα δημιουργήσει ε, και 25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, 7,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, το οποίο είναι ε, αναμενόμενο δεδομένο και των ποσοστών εκτέλεσης που έχουμε σήμερα και το πόσο ανθρώπων εργάζονται για την εκτέλεση αυτών των έργων. Και φυσικά μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων θα υπάρξουν και κάποιες ε, θέσεις εργασίας οι οποίες θα διαρκέσουν ε, για την Ήπερο ε, στο Δινεκές. Κυρίως λοιπόν θέλουμε να καλύψουμε διασυνοριακές πτυχές, γιατί αυτό το οποίο διαπιστώσαμε στα χρόνια της αξιολόγησης είναι ότι υπάρχουν εμβαλωματικά εθνικά δίκτυα, 27-28 εθνικά δίκτυα, τα οποία δεν συνδέονται και σίγουρα δεν συνδέονται διασυνοριακά. Και φυσικά αυτές ε, οι υποδομές ε, συνδέονται στενά και με τις ε, προσδοκίες για τις μεταφορές, διότι δεν θα πρέπει να συνδέσουμε διασυνοριακά τα δίκτυα αυτά, αλλά θα πρέπει να είναι και διαλειτουργικά για κάθε μέσο μεταφοράς, αλλά και συνδυασμένες μεταφορές. Πρόκειται λοιπόν για ε, πάρα πολύ σημαντικά πρότυπα, τα οποία πρέπει να υλοποιήσουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε συνολικά είναι το εξή. Καταρχά, επειδή πρόκειται για ένα διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, επομένω πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλε τι περιφέρειε. Και ε, γι' αυτό έχουμε και ένα συνολικό αλλά και ένα βασικό δίκτυο για να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε όλους. Ε, δεν πρόκειται απλώς ε, για ε, έργα αλλά και εναρμονισμό των προτύπων. Θέλουμε να έχουμε ε, ελεύθερη κυκλοφορία και ε, διασυνδεσιμότητα χωρίς ε, φραγμούς. Για παράδειγμα, θα γνωρίζετε ότι υπάρχουν 21 συστήματα ασφάλειας και προστασίας, τα οποία δεν είναι συμβατά. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και το ERTMS, το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε ένα αναρμοσμένο πρότυπο για τους σιδηροδρόμους. Και φυσικά θέλουμε να πάμε και πέραν αυτού, θέλουμε να έχουμε έξυπνες και καινοτόμες υποδομές και σταδιακά εισάγουμε και νέα πρότυπα, οποία καθορίζονται από τις πολιτικές μας. Για παράδειγμα, όσον αφορά το την πληροφορική και τις επικοινωνίες και την ψηφιοποίηση που είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά και εναλλακτικά καύσιμα. Και εδώ ερχόμαστε σε κάτι το οποίο επισημάνατε και εσείς ε, κυρία Πρόεδρε. Κάνουμε και αλλαγή από τα παραδοσιακά στα πιο ε, ε, ανανεώσιμα καύσιμα και φυσικά αυτό πρέπει να το εμβαθύνουμε και να το επιταχύνουμε. Δύο άλλα στιμία τα οποία πρέπει να αναφέρουμε είναι η κόμβη μεταφορών, γιατί εκεί γίνεται δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς όλοι οι λιμένες και τα αεροδρόμια, αλλά και οι δραματικοί σταθμοί ε, και φυσικά και αστική κόμβη, διότι εκεί τα διάφορα μέσα μεταφοράς συνδέονται. Αυτή είναι η βασική στόχη, αν θέλετε. Τώρα, οι προκλήσει που έχουμε ποιε είναι. Καταρχά για του στόχου υλοποίηση του 2030. Μπορούμε να έχουμε το βασικό δίκτυο μέχρι το 2030. Ε, καταρχάς, πρέπει να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει επαρκή προπολογισμό διαθέσιμο. Στο προηγούμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, συζητούσατε ακριβώ τον προπολογισμό. Εμεί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιε είναι οι ανάγκε, οι οποίε έχουν αξιολογηθεί πολλέ φορέ. τα βλέπετε στι διαφάνειε, 550 με 600 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030, αλλά φυσικά και ο προπολογισμό του 2020, ο οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και να επιταχύνουμε στι προτεραιότητέ μα. Το δεύτερο λοιπόν ε, σημείο είναι πολύ σημαντικό και θα είναι ουσιαστικό στοιχείο για την επόμενη αναθεώρηση των διευρωπαϊκών δικτύων. Θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε αυτέ τι επενδύσει για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και να αναβαθμίσουν τον εθνικό σχεδιασμά του. Στη χώρα σα, για παράδειγμα, κυρία Πρόεδρε, οι συζητήσει είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ε, για το θέμα. Βεβαίω, πρέπει να συνεχίσουμε και την εκτέλεση του δικτύου συνολικά δεν μπορούμε να είμαστε στάσιμοι σε κάποια σημεία και να μην υπάρχει συνέχεια. Η συνέχεια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει και να υπάρξει και επιτάχυνση. Ε, κάποια πράγματα τα οποία γινόντουσαν παραδοσιακά στο παρελθόν είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και να επιταχύνουμε προ τη βιωσιμότητα, προ εναλλακτικά κάστημα, ασφάλεια και ποιότητα υπηρεσιών. Και τέλο υπάρχει και το θέμα τη κινητοποίηση χρηματοδότηση, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τα κράτη-μέλη και από ε, δημόσιε και ιδιωτικέ πηγέ Προκειμένου να επιτευχθούν βεβαίω όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια, υπάρχουν οι Ευρωπαίοι συντονιστέ, τρει εξ αυτών είναι εδώ σήμερα, για να μα βοηθήσουν να καταλάβουμε ποιε είναι οι προκλήσει στον κάθε διάδρομο, τον κύριο Μπάλλα, ε, τον Ματία Γκρό και τον Κάρλο Σέκη. Και φυσικά οι συντονιστέ μπορούν να ε, έχουν ε, πρόσβαση στου ενδιαφερομένου πέραν των όσων μπορούν να κάνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εξωματούχοι, διότι είναι αυτοί οι οποίοι καταρτίζουν ένα σχέδιο εργασία με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ώστε όσα χρηματοδοτούνται μέσα των έργων να έχουν και κάποιο νόημα. Και φυσικά υπάρχει και συντονισμό όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ε, βλέπετε εδώ στη διαφάνεια λοιπόν τους ε, περιβόητους αυτούς εννέα διαδρόμους οι οποίοι καλύπτουν όλη την Ευρώπη και όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε υπάρχουν ε, δύο οριζόντια στοιχεία, το ERTMS και το Model TSE τα οποία συνδέονται με το Connecting Europe Facility. Ε, θα γίνει αναθεώρηση του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και ελπίζουμε να γίνουν ε, στη διάρκεια αυτής της θητείας αυτά όλα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζουμε και από την προηγούμενη αναθεώρηση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς ε, της Επιτροπής σας, διότι είναι ε, το βασικό στοιχείο για την εφαρμογή των προτύπων ε, για τους διαφορούς κόμβους αλλά και τις νέες πτυχές, τα καύσιμα, την πληροφορική και την επικοινωνία. Επομένως η Επιτροπή σας θα μπορέσει να επηρεάσει άμμοσα την πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων του μέλλοντος και Περιμένουμε και να ολοκληρωθεί μια μελέτη την άνοιξη του 2020. Έχει ε, γίνει και μια δημόσια διαβούλευση στη διάρκεια του θέρους και φυσικά θα συνεχίσουμε και τις διαβουλεύσεις από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο τον επόμενη χρονιά. Και αυτό θα ε, οδηγεί σε μια παρουσίαση το Μάιο του 2020 στις Διευρωπαϊκές ημέρες και από εκεί και πέρα θα έχουμε μια επίσημη πρόταση η οποία θα υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο εξάμεινο του 2021. Και αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα λοιπόν αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει βεβαίως ε, να δούμε και ε, πώς θα επιβεβαιωθεί όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όλα αυτά έχουν προβλεφθεί βάσει της ε, παρούσας θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, από εκεί και πέρα έχουμε να δούμε τι γίνεται με το σχεδιασμό του δικτύου. Είναι επαρκέ το δίκτυο, είναι αρκετά πυκνό, υπάρχουν συνδέσεις και με τρίτες χώρες όπως αναμένεται. Τα χαρακτηριστικά τώρα του δικτύου. Τα πρότυπα, όπως είπα, η διαλειτουργικότητα, ε, νέες κινητικότητα και φυσικά και στρατηγική στρατιωτική κινητικότητα και περιμένουμε ότι θα γίνει, για παράδειγμα, συζήτηση όσον αφορά κάποιε πτυχέ οι οποίε ε, συνδύονται με κόμβου, εναλλακτικά δίκτυα και ούτω καθεξής. Χρήση του δικτύου στη συνέχεια και τέλο εφαρμογή του δικτύου. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έθεσε και ο κύριο Μαρινέσκο, ο οποίο δεν είναι εδώ στην αίθουσα τώρα, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσουμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με την εκτέλεση των βασικών και συνολικών δικτύων. Ε, μπορούμε να τα επιτύχουμε μέχρι το 2030 όσα προβλέπουμε και και από εκεί και πέρα θα δούνε τι έχουμε να μας πείουν και οι Ευρωπαίοι συντονιστές και οι ενδιαφερόμενοι αλλά και εσείς. Δύο ακόμα ε, διαφάνειες για να ολοκληρώσω τη σύντομη παρουσίαση. Τώρα, το Connecting Europe Facility, κάτι το οποίο αναφέρθηκε και στην προηγούμενη, ε, στο προηγούμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, είναι πολύ σημαντικό για την υλοποίηση και την εφαρμογή της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και αυτό διότι ε, αντλούμε από αυτόν τον προπολογισμό για την εφαρμογή των ε, έργων αυτών και γιατί το ten και το ΣΕΦ ε, συστήθηκαν ταυτόχρονα και έχουν κοινού στόχους. Στην προηγούμενη εντολή έχουμε προχωρήσει με το ΣΕΦ 2 και έχουμε προχωρήσει και με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε μακρές διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Μαρινέσκου ήταν εκ των εισηγητών και ήσασταν και εσείς κυρία Πρόεδρε παρούσα μέχρι τις 4 τα ξημερώματα συζητούσαμε για τις ανάγκες ε, του προϋπολογισμού του νέου ΣΕΦ2. Και φυσικά Εκεί είναι σαφές ότι θα γίνει και μία αλλαγή προς ε, χρήση του προϋπολογισμού για πτυχές οι οποίες δεν είναι αμυγός ε, θέματα υποδομών, αλλά είναι ήπιες υποδομές όπως αποκαλούνται, δηλαδή εναλλακτικά καύσιμα, ασφάλεια, ε, πληροφορική και επικοινωνία κλπ. Αυτή τη στιγμή, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, έχουμε περίπου 85% τα οποία δαπανήθηκαν για το θέμα αυτό και στο νέο ΣΕΦ θα πάμε στο 60% και 40% για τις άλλες πτυχές. για τη συνογή είμαι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είμαστε στο 95% και θα προσπαθήσουμε να πάμε στο 85% με 15%. Αυξάνεται λοιπόν, τριπλασιάζεται ο προπολογισμό ε, στα θέματα αυτά και φυσικά υπάρχει και η ανάπτυξη των προϊόντων διετής χρήσης, ε, πολιτικής και στρατιωτικής, ε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν και υποδομές για στρατιωτικές μετακινήσεις. Ε, τώρα, όσον αφορά την Πράσινη Συμφωνία, το Connecting Europe Facility έχει ένα στόχο 60% δαπάνη που αφορά στόχους του κλίματος. Αυτός είναι ο υψηλότερο ε, στόχος που έχει υπάρξει ε, και έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό και η πτυχή των μεταφορών του Connecting Europe Facility, διότι ε, έχουμε ενέργεια, πληροφορική και μεταφορές. Ε, ε, οι μεταφορές είναι υψηλότερες από το 60% γιατί το βασικό σκέλος των επενδύσεων πηγαίνουν σε φιλικές προς το περιβάλλον δυνατότητες επικοινωνίας, τι προγράμματα έχουμε για κινητικότητα κλπ. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ καλό στόχο, τον οποίο μπορούμε να θέσουμε από κοινού. Και τελευταία διαφάνεια, κυρία Πρόεδρε, είναι μια ανοιχτή πρόταση, την οποία θέτω επιτάπητος ε, για, ε, για τον εξορθολογισμό των διευρωπαϊκών δικτύων. Ε, αυτός είναι ένας στόχος ε, ε για την προθεσμία του 2030. Μπορούμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά αρκετά γρήγορα και έχουμε καταλάβει ε, καλά πώς θα γίνει η εφαρμογή της πολιτικής, ε, την έχουν κατανοήσει οι πολίτες όσοι προωθούν τα θέματα ε, και πώς οδηγούν όλα αυτά στην εφαρμογή του κάθε στόχου. Η πρόταση αυτή είναι κάτι το οποίο απασχόλησε και την Επιτροπή σας. Υπάρχει ο συγητής, ο οποίος εξακολουθεί να είναι Ευρωβουλευτής Προσβλέπουμε λοιπόν και στην εφαρμογή όλων αυτών. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω οι συντονιστέ να ρίξουν φως ε, στα τρία συγκεκριμένα ε, προγράμματα που παρακολουθούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόιτερ, για αυτή τη γενική επισκόπηση, την παρουσίαση των πολύ γενικών στόχων. Καλό είναι να έχουμε στόχους και ακόμα καλύτερα να τους ε, υλοποιούμε. Όσον αφορά τα αντιευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, Μιλάμε για δίκτυα και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για τους ε, τρόπους αυτούς μεταφοράς που αφορούν τους επιβάτες, αλλά κυρίως τα εμπορεύματα. Να μην ξεχνάμε αυτήν την τεράστια πτυχή των μεταφορών το θέμα των εμπορευμάτων λοιπόν και όχι μόνο των επιβατών. Δεύτερον, που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι έχει αλλάξει εδώ η συμπεριφορά των Ευρωπαίων πολιτών. Σήμερα το θέμα των σιδηροδρομικών δικτύων αντιμετωπίζεται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, ένας Ευρωπαίος πολίτης θέλει να πάει από την μία πόλη στην άλλη και εσείς σαν συντονιστές θα πρέπει να λάβετε υπόψη όλα αυτά τα νέα δίκτυα όλους αυτούς τους νέους τρόπους μεταφορών, όπως παραδείγματος χάρη ανεκαλύπτω την Ευρώπη μέσω των σιδηροδρομικών μεταφορών και μέσω των ταξιδιών, παραδείγματος χάρη τη νύχτα, των νύχτερινών δρομολογίων. Θα σας δώσω όμως το λόγο στον καθένα από εσά για έξι λεπτά. Είμαι σήμερα πολύ γενναιόδορη και σας δίνω και δύο λεπτά παραπάνω στον καθένα. Κύριε Μπάλας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε και κύριοι, να σας συγχαρώ καταρχάς ε, τα νέα και τα παλιά μέλη αυτής της Επιτροπής, γιατί αντιμετωπίζετε μία από τις μεγαλύτερες ε, προκλήσεις του ευρωπαϊκού εγχειρήματος γιατί πρόκειται πραγματικά για την κυκλοφορία του αίματος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, οι μεταφορές. Εγώ ε, ε, είμαι ο γυρεότερος συντονιστής μεταξύ των συναδέλφων μου ε, και μάλιστα ήμουν παρόν όταν η Κομισιόν είχε κάνει ένα πολύ τολμηρό βήμα. Θα θυμάστε ότι στην αρχή υπήρχαν 30 έργα μεταφορών, ήταν ένα ολόκληρο μοσαϊκό αν θέλετε, αλλά το 2005 η Κομισιόν ανέλευε την τολμηρή πρωτοβουλία να καθορίσει πέντε έργα προτεραιότητε και να ζητήσει μάλιστα από πέντε πρώην επιτρόπου να γίνουν συντονιστέ αυτών των έργων. Εγώ είχα το προνόμιο να είμαι ένα από αυτού και ε, τότε ε, μάλιστα συντόνισα και τη συνδρομική σύνδεση του Παρισιού με την Πρατισλάβα μέσω Γερμανίας και Αυστρίας. Είχα τη χαρά λοιπόν να συμμετέχω σε όλη αυτή τη διαδικασία με την Γενική Διεύθυνση MOVE. Συνεργάστηκα με πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που ακριβώς ασχολήθηκαν με αυτήν τη νέα ε, φάση των ευρωπαϊκών μεταφορών που μας παρουσίασε και ο κύριος Ρόιτερ, ήταν ένα συνολικό αν θέλετε εγχείρημα, μια προσέγγιση συνολική, ολιστική που θα κάλυπτε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να γίνουν 9 διάδρομοι μαζί με τα συμπληρωματικά δίκτυα. Το νέο στοιχείο, το σημαντικότερο νέο στοιχείο ήταν η πολυτροπικότητα. Το πώς δηλαδή οι ισοδρομικές μεταφορές, οι οδικές μεταφορές, όλες οι άλλες, ε, όλα τα άλλα είδη μεταφορών θα μπορέσουν να συλλειτουργήσουν. Και εγώ λοιπόν ήμουν ε, συντονιστής για τον διάδρομο που συνδέει την Βόρεια Θάλασσα από την Σκοτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και κατεβαίνει προς τα κάτω κατά μήκο του Ηνωμένου Βασιλείου, την, ε, το, την Ιρλανδία, την Μπενελούξ έως και την ε, ηλιόλουστη Μασαλία. Βλέπετε εδώ αυτό το διάδρομο. Εκεί υπάρχουν πάρα πολύ πολλές μεταφορές, ε, πολλοί διάδρομοι μεταφορών, σειροδρομικοί, εσωτερικές πλωτές οδοί κτλ. Εργαστήκαμε λοιπόν μαζί με τους συναδέλφους μου σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τους εμπλεκόμενους φορούς και το βασικό στοιχείο των εργασιών μας ήταν αυτό το σχέδιο εργασιών που θέλαμε να καθορίσουμε, το οποίο έχει δημοσιευτεί κιόλα. Στον δικό μου διάδρομο αυτή τη στιγμή υλοποιούνται πάνω από 350 έργα σε έξι κράτη-μέλη που αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο ύψος επενδύσεων που είναι αναγκαίο να γίνουν και ανέρχονται σε πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή ο διάδρομος αυτός έχει λάβει 1,8 δισεκατομμύρια χρηματοδότηση από το ΣΕΦ για την υλοποίηση περίπου 85 έργων μικρής και μεγάλης έκτασης και πρόκειται για ένα συντελεστή πολλαπλασιασμού γιατί με αυτά τα 1,8 ε, δισεκατομμύρια καταφέραμε να κινητοποιήσουμε 5,2 ε, ε, ε, δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην απαλλαγή από τον άνθρακα και ε, προσπαθούμε να μεταφέρουμε τις εμπορευματικές μεταφορές από τους αυτοκινητοδρόμους στις εσωτερικές πλωτές οδούς και στους υδροδρόμους. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τρία βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Το πρώτο είναι το μεγαλύτερο δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών στην Ευρώπη, το Saint δίκτυο. Σενεσκό πολλές φορές στα γαλλικά το μπορείτε να το ακούσετε, που ε, συνδέει την ίδια λεκάνη μέσω των ε, ποταμών από την Βόρεια Γαλλία, μέσω Βελγίου, Ολλανδίας και πάει παραπέρα μέχρι το Ρήνο και τα λοιπά. Ε, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Το βασικό στοιχείο είναι η ε, σύνδεση 170 χιλιόμετρων στο κανάλι Σενόρ στη Γαλλία, τα οποία έλειπαν. Μόλις αυτό το κενό καλυφθεί, θα υπάρχουν ακόμα πιο εντατικές συνδέσεις και μεταφορές μεταξύ των περιοχών που σας ανέφερα. Καταφέραμε να κατακτήσουμε, να καταλήξουμε σε μια απόφαση ε, που αφορούσε τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα. Σιδηρόδρομοι. Οι σιδηρόδρομοι είναι ο μόνος τρόπος μεταφορών που συνδέει το ένα άκρο του διαδρόμου με το άλλο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Πέρα από το σύστημα TRTNS, το σύστημα σηματοδότησης και σήμανσης, η το μέτρο φόρτωση των τούνελ δυστυχώς δεν είναι ίσο σε, όλη την, όλο το μήκος του διαδρόμου αυτού και ε, γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να ε, διορθώσουμε αυτές τις ε, διαφορές που υπάρχουν για να μπορούν τα εμπορευματοκιβώτια να περνάνε καθόλου το μήκος του διαδρόμου. Και το τελευταίο στοιχείο που με αφορά και θέλω να, στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το Brexit. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο διάδρομο αυτόν και έχουμε καταφέρει μαζί με τον κύριο Σέκη να διοργανώσουμε ένα σεμινάριο στο Δουβλίνο για να αναλύσουμε τις μεταφορές από και προς την Ιρλανδία αλλά και ε, κατά μήκο της ε, ε γέφυρας ε, που είναι στην ουσία για τις μεταφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και βεβαίως έχουμε πάρει διάφορες περιπτώσεις, το σκληρό Brexit, έχουμε λάβει όλα τα, τα εχέγγυα ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ελπίζουμε όμως ότι το, αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα το οποίο θα, ε, ε, στο οποίο θα καταλήξουμε ε, θα αποσοβήσει τα χειρότερα. ξέρετε ότι το δημοψήφισμα δεν κατέληξε στην επιλογή να υπάρξει μια εναλλακτική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κατέληξε στο αποτέλεσμα της αποχώρησης. Πάντως ε, είμαι στη διάθεσή σας ε, και σας και όλων των συναδέλφων για να κάνουμε διμερείς διαβουλεύσεις αν το επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε σε αυτό το σχέδιο ε, και ιδιαίτερα υπό το φως των συνεπειών του Brexit. Θα δούμε τι θα γίνει εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Ο κύριος Σέκη. Έχετε το λόγο για τον διάδρομο του Ατλαντικού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας όσον αφορά τον Ατλαντικό διάδρομο, τον οποίο και ε, παρακολουθώ. Και βεβαίως προσβλέπω και εγώ όπως και όλοι οι συνάδελφοι σε μια πολύ γόνιμη συνεργασία τα επόμενα χρόνια μαζί σας. Ο Ατλαντικός διάδρομος περιλαμβάνει μια σειρά από διασυνορικές περιφέρειες που ε, χρειάστηκε είτε να χτιστούν είτε ε, πλήττονται από συμφόρηση και γι' αυτό χρειάστηκε ε, η οικοδόμηση σιδηροδρομικών δικτύων για να αποσυμφορηθεί η συμφόρηση στο, στους αυτοκινητοδρόμους. Ε, σας δίνω ως παράδειγμα τη σιδηροδρομική σύνδεση Γαλλίας-Ισπανίας για παράδειγμα εδώ στην ε, γραμμή Βιτόριο Μπορντό η οποία πρέπει να, να ε, ανασκευαστεί ή ε, ε, να δοθεί ένα από τα έργα με τα οποία ασχολούμαστε είναι η ενίσχυση των επιβατικών μεταφορών στην πλευρά της Γαλλίας και την οικοδόμηση, την κατασκευή γραμμών υψηλής ταχύτητας. Η Ισπανία θα, θα τελειώσει το έργο έως το σύνορά της με κάποια με κάποιες καθυστερήσεις, αλλά έως το τέλος του 2023 σε κάθε περίπτωση. Η Γαλλία, ωστόσο, ανέβαλε την κατασκευή των νέων γραμμών υψηλής ταχύτητάς της και γι' αυτό εγώ βρίσκομαι σε επαφή με το Γαλλικό Υπουργείο και τους εμπλικόμενους φορούς για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ε, μια ε, αναζωογόνηση της υπάρχουσας γραμμής από το Μπορντό έως τα γαλλοϊσπανικά σύνορα. Επίσης, αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην διασυνορική σύνδεση Πορτογαλίας-Ισπανίας, ε, ε, στη σύνδεση Λισαβόνας-Μαδρίτης. Πρέπει να, χτιστούν πρέπει να χτιστεί η σιδηροδρομική αυτή γραμμή στην Πορτογαλία από την αρχή και να ε, αναβαθμιστεί στην πλευρά της Ισπανίας. Βρισκόμαστε σε επαφή με τα δύο Υπουργεία για να υλοποιήσουμε αυτή τη σύνδεση έως το τέλος του 2030, δηλαδή στο τέλος της προγραμματικής μας περίοδου. Και ε, κατάφερα να αποσπάσω από την Κομισιόν μια εφαρμοστική απόφαση στο τέλος της περσινής χρονιάς για αυτήν την διασυνοριακή σύνδεση με την έγκριση των κρατών μελών που θεωρήθηκε ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ο Ατλαντικός διάδρομος επίσης έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του του εύρου των ε, σειροδρομικών γραμμών στην Ιβυρική Χερσόνησο. Θα πρέπει να αναβαθμιστούν όλες αυτές οι σειροδρομικές γραμμές προκειμένου να εναρμονιστούν με, τα, με το εύρος των ε, υπολείπων σειροδρομικών γραμμών στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά έχουμε και τις ε, ε, μεγάλες, μεγάλες αποστάσεις, τα, τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων που επίσης είναι μεγάλο ενδιαφέροντος για το δικό μας διάδρομο. Σύνδεση επίσης με το βασικό δίκτυο. Τον επόμενο μήνα ή τον παρεπόμενο, δεν το ξέρουμε ακόμα, θα γίνει μια συνάντηση στην Πορτογαλία για ε, της ε, ομάδας εργασίας για την περιφερειακή συνεργασία των Ατλαντικών πόλεων και δήμων και εκεί θα προσδιορίσουμε τις πλέον πιεστικές ανάγκες. Φυσικά το Brexit είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο ε, έχουμε προσπαθήσει να αντιμετωπίσουμε και ε, όπως είπε και ο συνάδελφος καθηγητής Μπάλας ε, πριν από λίγο, ο Ατλαντικός Διάδρομος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό ε, έχοντας κατά νου ότι από κάποιο σημείο και προς τα κάτω υπάρχουν, κάποιες, υπάρχουν πολλές δυνατότητες τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε στο μέλλον και από το Σαλαζάρ και πάνω βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Συνεχίζουμε λοιπόν τον ε, διάλογό μας με τους συνομιλητές μας προκειμένου να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε πιθανές λύσεις. Και όπως γνωρίζετε ίσως κάποιοι από εσάς, στην προτινόμενη αναθεώρηση του παρερτήματος 2 του κανονισμού για το ΣΕΦ, ένα από τα αντικείμενα που έχουν συζητηθεί είναι το πώς θα εντάξουμε ε, το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit ε, στα συστήματά μας είναι και αυτό κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει. Και αν μου επιτρέπετε, έχω προσπαθήσει να αντιμετωπίσω και άλλα προβλήματα οριζόντιας φύσης και συγκεκριμένα με τον συνάδελφο καθηγητή κύριο Κουρτ Μπόντεβικ προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε και να προσδιορίσουμε νέες ιδέες σε συνεργασία με όλους τους άλλους συντονιστές βεβαίως για να βελτιώσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας όχι μόνο ως προς το μέγεθός τους, αλλά και ως προς την καινοτομία για να προσελκύσουμε μεγαλύτερα ιδιωτικά κεφάλαια για να καλύψουμε τα χρηματοδοτικά μας κενά, όπως επισήμανε στην αρχή και ο κύριος Ρόιτερς. Μόλις έχουμε ολοκληρώσει αυτό το έγγραφο, το οποίο και θα θέσουμε στη διάθεσή σας τις επόμενες εβδομάδες για το πώς θα μπορέσουμε καλύτερα να προσαλκύσουμε και να ενσωματώσουμε ιδιωτικά κεφάλαια στη χρηματοδότηση των έργων μας. Έχουμε καταλήξει σε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσε ιδέες, τις οποίες βεβαίως βάζουμε στο τραπέζι της συζήτησης και τις οποίες θα θέλαμε να συζητήσουμε και μαζί σας. Είναι πολύ ε, σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή να τα συζητήσουμε όλα αυτά και μαζί σας. Σας ευχαριστώ κύριε Σέκη. Είστε πάρα πολύ φιλόδοξος βλέπω. Μας μιλάτε για την γραμμή Λισαβόνα Μαδρίτη. Λέτε σε δέκα χρόνια. Μα τι λέτε. Το 30 είναι σε 10 χρόνια. Όλες αυτές οι διαστηνές πρέπει να γίνουν με μεγάλα βήματα και με ταχύτατους ρυθμούς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε στο 2030 η Επιτροπή μας Βεβαίως κοιτάει το θέμα της χρηματοδότησης, αλλά κυρίως κοιτάει το θέμα των προτεραιοτήτων. Και αυτό που μας ζητάνε σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πολύ συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Αν θέλει κάποιος να πάει από τη μία πρωτεύουσα στην άλλη, δεν μπορεί να περιμένει 10 χρόνια. Και αυτή είναι για μας η πρόκληση ήταν ένας από τους στόχους μας το άνοιγμα του διαδρόμου του Ατλαντικού. Κύριε Ρικέ, είστε στις διαπραγματεύσεις για το Brexit. Θα πρέπει να ανοίξει λοιπόν αυτός ο διάδρομος του Ατλαντικού, να υπάρξει ένα νέο δίκτυο το οποίο να συμπεριλαμβάνει και τους ε, αυτοκινητόδρομους όπως ε, τους ονομάζουμε, τους δρόμους και τις θαλάσσιες διαδρομές. Κύριε Κρός, Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που μπορώ σήμερα να ξαναδώ τα παλιά μέλη της Επιτροπής, να συναντήσω τα καινούρια. Θέλετε κάτι το συγκεκριμένο, είπατε, αυτά αποτελέσματα. Θα σας δώσω λοιπόν απλά και απτά αποτελέσματα. Ε, έχω προετοιμάσει μια ομιλία με διαφάνειες, ελπίζω να μοιραστεί σε όλους. Εγώ όμως θα σας μιλήσω για τους πολυτροπικούς διαλόγους, 5.800 ε, χιλιόμετρα και μεγάλης γεωστρατηγικής ε, σημασίας είναι ο διάδρομος ο οποίος ονομάζεται Ανατολικός, Ανατολική Μεσόγειος από την Βόρεια Ευρώπη στην Ελλάδα, στα λιμάνια της Ελλάδας, από τη Γερμανία μέχρι τα λιμάνια της ε, Νότιας Ελλάδας. Ένα μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πολύ συγκεκριμένες προκλήσεις. Η προσέγγιση μας είναι τεχνική. Θέλουμε πραγματικά τεχνικά κριτήρια και αυτό που κάναμε για τους συγκεκριμένους αυτούς διαδρόμους επιλέξαμε κυρίως τις εσωτερικές πλωτές οδούς καθώς και το σιδηρόδρομο. Αν πάρετε παραδείγματο χάρη το τρένο βόρεια για να πάτε νότια πρέπει να αλλάξετε έξι φορές τις μηχανές των τρένων. Πρέπει να αλλάξετε το μήκος, αν θέλετε, των σιδηροτροχιών. Πρέπει να αλλάξετε το συγκεκριμένο βάρος ε, το αξονικό, διαφορετικές ε, τεχνικές προδιαγραφές, διαφορετική ταχύτητα. Αν κοιτάξετε αυτόν το χάρτη θα διαπιστώσετε τις τεράστιες διαφορές που συνεχίζουν να υπάρχουν σε αυτούς τους διαδρόμους. 460 πολύ σημαντικά σχέδια έχουν υποβληθεί και προς το παρόν 94 υλοποιούνται. 94 με έναν προϋπολογισμό πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε προτεραιότητα και το υπογραμμίζω αυτό με 85% επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και αυτό είναι κάτι που για μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Αν κοιτάξετε την κατανομή αυτών των ε, προγραμμάτων, υπάρχουν διασυνοριακές επενδύσεις, υπάρχουν τα λεγόμενα missing links, δηλαδή οι διασυνδέσεις που δεν υπάρχουν και μέχρι το 2023 πιστεύουμε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει αυτά τα 94 προγράμματα που έχουν ξεκινήσει, ηλιοποιώντας βεβαίως και καινούρια. Θέλουμε να υπάρξει συνέχεια στις προσπάθειες και επαναλαμβάνω ότι το συνολικό πλαίσιο χρηματοδότησης μέχρι το 2030 θα συμπεριλάβει 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εσωτερικές ε, πλωτές ε, οδοί, ο στη Βόρεια Γερμανία και η διασύνδεση με έναν πολύ τεχνικό και έντονο διάλογο μεταξύ των Γερμανών και της Δημοκρατίας της Τσεχίας με τον Gesamtkonzert Elbe και νέες προτάσεις για να δημιουργηθεί ίσως ε, πολύ σύντομα νέες διασυνδέσεις στην περιοχή του Έλβα. Επίσης ε, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες διπλωματικές, πολιτικές και η συνεργασία μεταξύ της Γερμανίας και της Δημοκρατίας της ε, ε, Τσεχίας ήταν εξαιρετική και έχει προχωρήσει πολύ σημαντικά. Δρέσδη, Πράγα, εδώ θέλουμε να ξεπεράσουμε την συμφόρηση και τα διέξοδα, τα λεγόμενα bottlenecks, Μεταξύ Πράγας λοιπόν και Δρέσδης υπάρχει τεράστια συμφόρηση κυκλοφοριακή και στο οδικό δίκτυο αλλά και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και αν κανείς δει ακριβώς τη συχνότητα αυτών των ε, διαδρομών, στηρίζουμε το shift to rail, δηλαδή πώς θα μεταφέρουμε τις ε, διαδρομές αυτές όλο περισσότερο από το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων, από το οδικό δίκτυο προς τον σιδηρόδρομο περιληπτικά. Θέλω να σας πω ποιες είναι οι σημαντικές προκλήσεις αυτού του διαδρόμου. Η χρηματοδότηση. Ένα τεράστιο θέμα, μια μεγάλη πρόκληση και πιστεύω ότι εδώ το ΣΕΦ 2 θα είναι μεγάλη στήριξη για μας. Δεύτερον, το θέμα των διαρθρωτικών κονδυλίων. Υπάρχουν περιοχές που χρηματοδοτούν σε κάποιες περιοχές χρηματοδοτούνται όλες αυτές οι υποδομές των μεταφορών πολύ περισσότερο από τα διαρθρωτικά κονδύλια από ό,τι από το ΣΕΦ. Υπάρχουν όμω και άλλες πολύ σημαντικέ προκλήσεις, τις οποίες πολλέ φορές δεν λαμβάνουμε αρκετά σοβαρά υπόψη. Συνέπειε στην ανάπτυξη, Συνέπειε για το κλίμα, και όσον αφορά την, τον σχεδιασμό του διαδρόμου μας, εμείς έχουμε κάνει ειδικέ μελέτες αντικτύπου και για το κλίμα αλλά και για την ανάπτυξη. Περιβάλλον λοιπόν και ανάπτυξη και η μη υλοποίηση, η μη εφαρμογή κάποιων συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων και κανονιστικών μέτρων έχει τεράστιο αντίκτυπο. Υπάρχουν όμως κράτη, και το ξέρουμε σήμερα, που δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα σχέδια. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις χώρες που βρίσκονται στον, ε, στον της συνοχής. Και σε άλλες χώρες υπάρχουν ελλείψεις και αδυναμίες στις εθνικές δομές, έτσι ώστε να γίνει σωστή διαχείριση αυτών των ε, σχεδίων. Και μια άλλη παρατήρηση. Πολλές φορές επενδύουμε ένα δισεκατομμύριο για να κερδίσουμε μία ώρα. Και όπως σας είπα, κυρία Πρόεδρε, και έχετε δίκιο, στον διάδρομο μεταφοράς εμπορευμάτων υπάρχουν σήμερα στις ε, παραμεθόριες περιοχές και στις διεθνωριακές ε, περιοχές συγκεκριμένες δυσκολίες, καθυστερήσεις. Πολλές φορές υπάρχουν πάνω από 30 ώρες αναμονή και καθυστέρηση στις περιοχές αυτές. Και εδώ μιλάμε για bottlenecks, εδώ μιλάμε για συμφόρηση, υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας, υπάρχουν όμως προβλήματα και ανταλλαγής πληροφοριών και υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες οι οποίες μπορούν να ξεπεραστούν. Ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν περιοχές που περιμένουμε έναν αστυνομικό έλεγχο για τρεις ώρες. Περιμένουμε την αλλαγή μιας ε, μηχανής του τρένου για τέσσερις ώρες. Όλα αυτά είναι θέμα συνεννόησης, είναι θέματα που μπορεί να ξεπεραστούν και να μην περιμένουν 30 ώρες, αλλά δύο. Σήμερα έχουμε 240 πρωτοβουλίες τις οποίες προσπαθούμε να υλοποιήσουμε για να βελτιώσουμε πολύ συγκεκριμένα την ε, κατάσταση αυτή. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της χρηματοδότησης, αλλά υπάρχει και το θέμα της συνεργασίας και της υιοθέτηση των βέλτιστων λύσεων. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλους τους τρόπους μεταφορών, κυρίως όμως το σιδηρόδρομο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκρός, λέει Πρόεδρος. Το θέμα είναι οι καθυστερήσεις. Έχετε δίκιο. Σε κάποιες περιοχές και όχι μόνο διασυνοριακές. Εμείς όταν πήγαμε στην Ελλάδα και είχαμε την τιμή να έχουμε την κυρία Κουντουρά στον πλευρό μας, η οποία ήταν τότε υπουργό Τουρισμού. Οι καθυστερήσει στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων, ήταν δύσκολο να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να περάσει από μία νοοτροπία οδικών μεταφορών από τη μία μέρα στην άλλη στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζεται θάρρος. Θα ξεκινήσουμε όμως αμέσως τη συζήτηση. Κυρία Τάλερ, καλημέρα σας. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ ε, τους συντονιστές ε, για τις παρουσιάσεις τους. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ολόψυχα ότι η ολοκλήρωση των δικτύων θα μειώσει αρκετές πιέσεις στα υφιστάμενα δίκτυα και θα είναι φυσικά και ένα εξοχό επίτευγμα όταν θα ολοκληρωθεί. Ωστόσο, στη δική μου την περιφέρεια, εγώ είμαι από το Τυρόλο, θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά τη ε, χρονολογικό συντονισμό των διασυνοριακών κατασκευών. Υποτίθεται ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα συνδέσουν τις οικονομίες μας και θα δώσουν όθεση στις διασυνοριακές σχέσεις. Αλλά χωρίς ε, εποπτεία από πάνω προς τα κάτω, οι διάφορες περιφέρειες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιταχύνουν τις ε, εξελίξεις ε, και την κατασκευή πέραν των συνόρων τους. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι πώς σκοπεύετε να εξορθολογήσετε το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων χωρών ώστε να αποφύγουμε καθυστερήσεις. Και η δεύτερη ερώτηση είναι τι γίνεται με τα οικονομικά ωφέλη και το κόστος. Όπως αναφέρεται και στο σημείο το ενημερωτικό, ε, αναφέρεται ότι υπάρχουν τεράστια ωφέλη για τις χώρες εάν εκτελέσουν σωστά τα έργα, αλλά Εάν μια άλλη χώρα καθυστερήσει την ε, κατασκευή του δικού τους του σκέλους, η χρηματοδότηση της ε, άλλης χώρας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, όσο αποτελεσματικά τουλάχιστον όσο προβλέπεται. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ραμόν Δίας, Μπαουσάς Δίας, ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το ευρωπαϊκό όνειρο δημιουργήθηκε πριν από 50 χρόνια με την ε, υπόσχευση να δοθεί ελευθερία στους πολίτες. Δύο μορφές ελευθερίες ε, στην ουσία. Προσωπική ελευθερία με τη δυνατότητα να ζει κάποιο, να ταξιδεύει και να εργάζεται και να σπουδάζει οπουδήποτε, αλλά και με οικονομικέ δυνατότητα, ώσπου οι πολίτε αλλά και οι επιχειρήσει θα μπορούσαν να ε, εμπορεύονται ε, τα αγαθά και τι υπηρεσίε του παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα, αλλά ε, δεν είναι αλήθεια ότι έχουν ιδρυωθεί με τον ίδιο τρόπο σε όλε τι χώρε και σε όλε τι πλευρέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την περίπτωση, γιατί το ανέφεραν και οι συντονιστέ τη παρουσιάση Στι ε, στις περιφερειακές χώρες. Ε, χώρες ε, στις οποίες μπορούμε να ρωτήσουμε τι γίνεται όταν κράτη-μέλη όπως η Ισπανία, όπως η Πορτογαλία, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα ή και η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν διαθέτουν απαραίτητες υποδομές για να μπορέσουν να καλύψουν αυτή την βασική ελευθερία που πολύ σωστά είπε και η Πρόεδρος, δεν είναι μόνο η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων αλλά και εμπορευμάτων, αγαθών υπ' αυτήν την έννοια, αυτό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους που έχουμε όλοι ως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δόθηκαν κάποια παραδείγματα από τους συντονιστές, αλλά επιτρέψτε μου να σας δώσω κι εγώ ένα παράδειγμα ε, για την Ισπανία. Δεν θα αναφερθώ ε, στην περιφέρεια στην οποία είμαι πρόεδρος, δεν θα ήταν σωστό, αλλά σε μια περιφέρεια πολύ σημαντική της ε, Μεσογείου, της περιοχής της Μούρθια, η οποία είναι λεγόμενη πόρτα της Ευρώπης. Η Μούρθια είναι μια περιοχή πάρα πολύ ανταγωνιστική, έχει εξαγωγές και παραγωγή, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να έχει αυτή την ανταγωνιστικότητα όπως οι υπόλοιπε περιοχές της Ευρώπης, ακριβώς γιατί δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές. Και εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει, και μιλάω ως συντονιστό ε, στην ομάδα στην οποία ανήκω, του Renew Europe, εμείς είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, ε, να υπάρχουν αυτοί οι διάδρομοι, γιατί είναι ζωτικοί άξονες. Και αυτό όχι μόνο για τις περιφερειακές χώρε μέλη, αλλά και για τις περιοχές τους, όπως τη Μούρθια, την Πελοπόννησο, τη Σικελία. Ο, κάθε χώρα έχει τις περιοχές της και ε, ε, θα έπρεπε όλοι να διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες. Νομίζω ότι αυτό είναι ο βασικός στόχος, είναι ο πιο σημαντικός στόχος ε, όλων όσων είμαστε εδώ και Φυσικά εμείς θα πρέπει να ενισχύσουμε όλες αυτές τις πτυχές και θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Και εδώ μιλάω όχι μόνο ως συντονιστής ε, της ομάδας μου, αλλά και ως ε, πολίτης αυτών των περιφερειακών χωρών που συμμετέχουν και στην ομάδα μου. Η ερώτηση σου είναι μία ε, πολύ συγκεκριμένη και το σχολίασε και η πρόεδρος προηγουμένως. Πότε δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε πολύ. Πότε λοιπόν αυτές οι περιφερειακές χώρες, αυτές οι περιφέρειες των ε, περιφερειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες να εκμεταλλευτούν αυτή την ευρωπαϊκή έννοια της ελευθερίας της μετακίνησης, ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, ατόμων και υπηρεσιών. Διότι αν δεν γίνει και αν δεν υπάρχουν προ... συγκεκριμένες προθεσμίες, ε, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας, θα είναι ένα στόχος πάρα πολύ ε, δόκιμος μεν, αλλά που δεν θα μπορεί πολύ εύκολα να επιτευχθεί. Ε, εδώ είμαστε στη, στη διάθεσή σας για να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε, αλλά θα πρέπει ε, στο τέλος να σκεφτούμε τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κόφη, το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους ε, καλή επιστροφή. Θα θέσω το ερώτημά μου στα γερμανικά. Έχω ένα ερώτημα για τον προπολογισμό και για τη χρηματοδότηση προς τους συντονιστές. Ως πράσινοι φυσικά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να σας υποστηρίξουμε ε, στον στόχο που έχετε θέσει να απαλλαγούμε στην Ευρώπη στις μεταφορές μας από τον ένθρακα και για να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων πολλών. Αλλά δεν κατάλαβα, ο προπολογισμό σας με ποιον ακριβώς και τα διάφορα στοιχεία του, τα διάφορα τμήματά του, πώς ακριβώς αλληλεπιδρούν, πώς ε, συλλειτουργούν αν θέλετε. Γιατί για μας είναι ξεκάθαρο ότι τα διασυνοριακά έργα που είναι και ο πυρήνας του έργου σας ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά και όταν, όπως μας είπατε εσείς, ότι υποχρηματοδοτούνται αυτά τα έργα, προφανώς δεν μπορούμε να επιτύχουμε, να επιτύχουμε όλοι μαζί και εμείς και εσείς τους στόχους που έχουμε θέσει. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πώς θα μπορούσαμε εμείς από την πλευρά της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σας υποστηρίξουμε στην ενίσχυση της χρηματοδότησης αυτών των διασυνοριακών έργων, πώς θα ενισχύσουμε τον σιδηρόδρομο, το σιδηρόδρομο, ιδίως τα νυχτερινά βαγόνια, γιατί Επιτακτικά, επιτακτική είναι πλέον η ανάγκη να εξευρεθούν εναλλακτικέ ιδίω όσον αφορά την αεροπορία. Ε, αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Αφορά τον προπολογισμό και τη χρηματοδότηση το ερώτημά μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τσίλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που επανήλθαμε εδώ. Σας ευχαριστώ όλους τους συντονιστές για τις παρουσιάσεις. Έχω δύο ερωτήσεις, μία προς τον κύριο Ρόιτερς, όσον αφορά τα θέματα της χρηματοδότησης cash flow και όσον αφορά την Connecting Euro Facility 1 και 2. Από το 1, το SEF 1, περιμένετε ακόμα χρηματοδότηση για τη συνοχή. 19-20, τη χρηματοδότηση για τη χρονιά μέχρι το 20. Κατόπιν Μπορεί να υπάρξουν και θέματα με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και βεβαίως εδώ μπορεί να δημιουργηθούν ε, δυσκολίες cash flow για τις χρονιές 21-22. Εάν δεν ξεκινήσουν για το κεντρικό δίκτυο, κάποια προγράμματα, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές ε, αυτές περιοχές που συνεχίζουν και υπάρχουν προβλήματα, προβλήματα που υπάρχουν εδώ και χρόνια και τα οποία θα συνεχίσουν να τα αντιμετωπίζουμε. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς ποια είναι η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συνοχή, διότι μία με το καλό, μία με το κακό βλέπω εδώ να προχωρούμε, να ε, κινητοποιούμε τα διάφορα προγράμματα, πώς θα τα κινητοποιήσουμε με έναν σημαντικό τρόπο από εδώ και πέρα. Άκουσα τους συναδέλφους. Εσείς όμως, όσον αφορά το τέλος της επόμενης περίοδου, το 2027, και τρία χρόνια πριν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων το 2030 του κεντρικού δικτύου, περιμένετε να έχουν ολοκληρωθεί ή σχεδόν ολοκληρωθεί τα ε, βασικά αυτά σχέδια, εσείς σαν συντονιστής, ανησυχείτε για κάποια από αυτά ή όχι. Ευχαριστώ πολύ, Ρόμπερ. Η κυρία Κουντουρά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συντονιστές για το έργο τους και για τη σημερινή ενημέρωση. Στην Επιτροπή μας ανάμεσα στις βασικές θεματικές που μας απασχολούν είναι η διείσδυση των σιδηροδρόμων και οι συνδυασμένες μεταφορές όσο με δύο σημαντικούς στόχους να γίνουν οι μεταφορές συμβατές με τους κλιματικούς στόχους και παράλληλα να ανοίξουν νέοι διάδρομοι δημιουργώντας τις βασικές προϋποθέσεις για ανάπτυξη, κυρίως σε περιοχές με ελλειπές δίκτυο υποδομών. Ειδικά για το δεύτερο σημείο, θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσά, κύριε Γκρός, καθώς η περιοχή για την οποία είστε υπεύθυνο είναι ο διάδρομος που ονομάζεται Ανατολική Μεσόγειος και φυσικά ε, είναι ο διάδρομος που ξεκινάει από τα Βαλκάνια και κατεβαίνει κάτω μέχρι την Ελλάδα. Και είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα στην Ευρώπη. Γνωρίζετε καλά ότι στην Ελλάδα οι σιδηροδρομικές μεταφορές αποτελούν, όπως ανέφερε και η κυρία Πρόεδρος που επισκέφθηκε πέρυσι με την Επιτροπή την Ελλάδα, ένα πολύ μικρό ποσοστό κυρίως των παθογενειών του παρελθόντος και διαχρονική ίσως έλλειψη πολιτικής βούλησης. Ωστόσο, τα τέσσερα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές προσπάθειες να ολοκληρωθούν έργα που θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί πάνω από μία δεκαετία πριν. Και για πρώτη φορά μάλιστα εκπονήθηκε στρατηγικό σχέδιο για τις μεταφορές με ορίζοντα το 2037. Στην επίσκεψή σας στη χώρα μας είχατε την ευκαιρία και εσείς ο ίδιος να το διαπιστώσετε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το διάστημα μπήκαν επίσης τα θεμέλια για τη δημιουργία του νέου διατροπικού διαδρόμου πανευρωπαϊκής σημασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, ο οποίος θα βασίζεται στη σιδηροδρομική σύνδεση των κομβικών λιμένων των δύο χωρών Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Μπουργάς Βάρνα Ρούσε με απότερο στόχο την παράκαμψη των στενών του Βοσπόρου όπου υφίσταται και υψηλός κορεσμός. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω επειδή μας ενημερώσατε ότι τα 94 σχέδια που ήδη υλοποιούνται με δύο δις μέχρι το 2023 θεωρείται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί αλλά έχουν κατατεθεί 460 σχέδια τι πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις των εμπλεκόμενων κρατών για να προχωρήσει ο διάδρομος με την ίδια δυναμική των τελευταίων χρόνων αλλά και ποια έργα θεωρείται ότι πρέπει να προχωρήσουν κατά προτεραιότητα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες ώστε να διατηρηθεί αυτή η δυναμική των τελευταίων ετών και να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε άμεσα. Merci Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να στραφώ προς τον Χάρετ και την Επιτροπή. Όσον αφορά τα μεγάλα δίκτυα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εδώ και 25 χρόνια δημιουργούν εργαλεία, δημιουργούν διευρωπαϊκά δίκτυα. Έχουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουμε τα περιφερειακά ταμεία, παραδείγματο χάρη, που ήταν πριν, προϋπήρχαν του Connecting Europe Facility. Και βεβαίως αυτό θα αντικατασταθεί σήμερα με το Invest Europe. Δημιουργούμε οργανισμούς, δημιουργούμε υπηρεσίες προτυποποίησης και όπως είπε πολύ σωστά ο Ματιό, τι νόημα έχει να δημιουργούμε ένα ενιαίο δίκτυο σιδηροδρομικό από τη στιγμή που τα τρένα αυτά καθεαυτά δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, σταματούν στα σύνορα, περιμένουν αλλαγή, ε, προσαρμογή και η ροή της κυκλοφορίας δεν είναι απρόσκοπτη. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι ότι πρώτον θα έπρεπε για τα δίκτυα να βαθμολογούμε τις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη για το περιβάλλον. Οικονομική βαθμολόγηση, κοινωνική βαθμολόγηση, αλλά και βαθμολόγηση όσον αφορά τα κοινά πρότυπα και την συμβατικότητα όλων αυτών των δομών και όλου αυτού του εξοπλισμού. Λειτουργούν διάφορα εργαλεία και βλέπουμε ότι η δυσκολία είναι να συνεπάρξει εθνική, περιφερειακή και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση η οποία να στοχεύει προς την ίδια κατεύθυνση. Γιατί κανείς μπορεί να κοιτάξει και το Invest Europe και το ΣΕΦ, αλλά και περιφερειακές και εθνικές πηγές χρηματοδότησης για τη στήριξη αυτών των έργων. Περιμένουμε το, τις εργασίες του Πρόεδρου Σέκη, ο οποίος εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως μία χρηματοδότηση οριζόντια, η οποία θα πρέπει να στηρίξει τα έργα αυτά. Εγώ είμαι εισηγητής για την οδηγία όσον αφορά την απλοποίηση την διοικητική των smart διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, γιατί στα μεγάλα δίκτυα, ακόμα κι αν όλοι συμφωνούν, όταν θελήσουμε να τα λειτουργήσουμε, υπάρχουν διάφορες φάσεις διοικητικέ, οι οποίες φτάνουν τα 8 χρόνια. Όταν όλοι συμφωνούν, όταν υπάρχει χρηματοδότηση, παρόλα αυτά περιμένουμε 8 χρόνια. Ακόμα και στο, εσωτερικό μίας χώρας δεν μπορούμε να οργανώσουμε τη λειτουργία. Καταλαβαίνετε όταν υπάρχουν και διευρωπαϊκές και διασυνοριακές ε, λειτουργίε, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσουν αυτά τα δίκτυα. Χρειάζεται λοιπόν όσον αφορά τα πρότυπα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση και όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες, απλοποίηση και νέα όθηση. Θα σας ακούσουμε λοιπόν και θα περιμένουμε τις προτάσεις σας και περιμένοντας όλα αυτά που θα μας πείτε θέλω να κάνω δύο ερωτήσει στους συντονιστές των δικτύων. Ματιέ, το τοπίο, το πολιτικό τοπίο στο νότιο τμήμα του δικτύου φαίνεται ότι αλλάζει. Οι σχέσεις της Μακεδονίας με την Ελλάδα έχουν αλλάξει πολύ, έχουν βελτιωθεί ευτυχώς. Η πολιτική στα Βαλκάνια είναι εν κινήσει και στην περιοχή αυτή γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες και τα νέα δεδομένα. Πώς αναλύεται αυτά τα νέα γεγονότα και αυτά τα νέα δεδομένα όσον αφορά την πρόοδο των ε, προγραμμάτων. Και στρέφομαι και προς τον κύριο Σέκη όσον αφορά τον Ατλαντικό διάδρομο. Μιλάμε ακόμα σήμερα για τον απεγκλωβισμό της Ιβηρικής Χερσονήσου και αναφερόμαστε στο πρόβλημα των πυρηναίων, στο εμπόδιο των πυρηναίων. Μα από τις δύο πλευρές υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα και θα έπρεπε επιτέλους η Ευρώπη να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ατλαντικός λοιπόν διάδρομος και το πρόβλημα των Πυρηναίων. Επίσης, σε αυτόν τον Ατλαντικό διάλογο υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης από δυσμάς προς Ανατολάς. Παραδείγματος χάριν, η Βρετάνοι, η οποία δεν είναι χαρακτηρισμένη σαν εξόχως περιφερειακή και απομακρυσμένη περιοχή, βρίσκεται στη Γαλλία και έχει πρόβλημα. Τι θα αλλάξει λοιπόν με το Brexit? Τα προβλήματα και οι συνθήκες θα αλλάξουν, αλλά παραδείγματος χάρη η Ατλαντική ακτή της Γαλλίας και όλη η δυτική περιοχή της Γαλλίας από την περιοχή Λαροσέλ μέχρι τα βόρεια της Βρετάνης που δεν συμπεριλαμβάνονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα και θα πρέπει και αυτές να απεγκλωβιστούν. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Ντέλη έχει το λόγο. Δεν είναι εξαδερφός μου ο κύριος Ντέλη, σας το υπενθυμίζω. Merci, Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα κυρίως στους κύριους Reuters και Gross. Γιατί αναφέρθηκαν σε ένα ζήτημα που θεωρώ πολύ σημαντικό, τη διεύρυνση των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Αν θυμάμαι σωστά, πριν από κάποιους μήνες, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δώσαμε την έγκρισή μας στη συμφωνία για τη δημιουργία της κοινότητας μεταφορών με τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Βασικός στόχος αυτής της κοινότητας είναι ο σχεδιασμός στον τομέα των υποδομών, ε, αποσυμφόρηση, διασυνδεσιμότητα κτλ. κτλ ιδίως η διασυνοριακή. Βλέπετε εσείς ως Κομισιόν, που συμμετέχετε βέβαια σε αυτή τη διαδικασία ενεργότατα, βλέπετε να έχει αποφέρει καθόλου καρπούς η συνεργασία στο πλαίσιο αυτής της κοινότητας. Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε διδάγματα από άλλες περιοχές σε αυτήν την συγκεκριμένη περιοχή. Πώς θα μπορούσαμε να την καταστήσουμε πιο συμβατή, αν θέλετε, με το δίκτυο TNT. Γιατί άμα δείτε τις ειδήσει που μας έρχονται από αυτές τις χώρες, θα δείτε ότι ε, υλοποιούνται μια σειρά από πολύ μεγάλα έργα υποδομών εκεί και με ενδιαφέρει να μάθω αν αυτά κατά τη δική σας αξιολόγηση είναι συμβατά με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός. Αφετέρου, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει στην προώθηση αυτών των έργων. Και τέλος, όλες αυτές οι εξελίξεις που υπάρχουν θα ληφθούν υπόψη στην συνολική αξιολόγηση των, των δικτύων TNT που εσείς θα διενεργήσετε ως το τέλος του 2023 ή και νωρίτερα. Γιατί νομίζω ότι στόχος και σκοπός μας θα πρέπει να είναι να προωθείτε η διασύνδεση όλης της Ευρωπαϊκής Υπήρου και να καλυφθούν αυτά τα κενά που υπάρχουν στις διασυνδέσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ κυρία Μπλιμπάου Βαραντίκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ε, ελπίζω να ξεκουραστήκατε σε αυτές τις διακοπές γιατί η δουλειά που μας περιμένει είναι τεράστια όπως ακούμε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με τα λόγια του κυρίου Ρόιτερ, ο οποίος έλεγε ότι οι χώρες πρέπει να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στα διευρωπαϊκά σχέδια. Και αυτό είναι αυτό το οποίο μας λείπει. Μπορούμε να συζητούμε για διοικητικά προβλήματα αλλά στην ουσία αυτό συζητούμε τα τελευταία χρόνια και αναφέρομαι στα τελευταία χρόνια διότι για να μην μιλήσω για το 1994, όταν καθορίστηκαν τα σχέδια προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2003 έγινε αναθεώρηση των ε, προγραμμάτων και ε, επικυρώσαμε και πάλι ότι πρόκειται για απαραίτητα έργα για να μπορέσουμε καταρχάς να αντιμετωπίσουμε την κυκλοφοριακή συμφέρεση, να μπορέσουμε να έχουμε ε, δυνατότητα κυκλοφορίας ατόμων και εμπορευμάτων, να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα. Και τι συνέβη, αυτό το οποίο συνέβη είναι αυτό το οποίο μας έλεγε η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ότι τα κράτη-μέλη δεν έκαναν αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση των ε, χρηματοδοτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν και των ε, ε, χρηματοδοτικών πόρων από το δικό τους προϋπολογισμό, γιατί δεν έδωσαν προτεραιότητα σε αυτά τα έργα. Και τι συνέβη σε πολλές χώρες, κατασκευάστηκαν τμήματα των ε, σχεδίων προτεραιότητας ε, και ε, από εκεί και πέρα έχουν παραλύσει για αρκετά χρόνια. Και όχι μόνο ξοδέψαμε χρήματα, αλλά χάνουμε συνέχεια χρήματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σαφές και θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι τι μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας, ώστε να απαιτήσουμε με σοβαρό τρόπο για άλλη μια φορά από τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν αυτά τα προγράμματα. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος και υπάρχουν εκθέσεις και υπάρχουν και στοιχεία. Δεύτερον, το 2013, μετά από την αναθεώρηση, έγινε αναθεώρηση και του κανονισμού. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα του συντονιστέ για την πολύ πολύ πλοκή διπλωματική και διακριτική δουλειά που κάνουν όταν δεν μα ε, ε, λένε όλη την αλήθεια στι ερωτήσει που, ερωτήσεις που του κάνουμε για τη συμπεριφορά των κρατών μελών. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σα. Αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω επίση ότι σήμερα, με τη βελτίωση τη οικονομία από το 2020, από το 2008 και μετά, συγγνώμη, στα διάφορα διάφορα κράτη-μέλη, ε, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε ε, προβλήματα κυκλοφοριακή συμφέρουση, τα οποία ξοδεύουμε το 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ε, μπορούμε να το βελτιώσουμε. Δεν αντιδρούμε όμως και αυτό δεν είναι ευθύνη των θεσμικών οργάνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω πραγματικά ότι σοβαρά πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ε, ανασκουμποθούν γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεύτερον, είμαι πάρα πολύ ανήσυχη για το σχέδιο για τον Ατλαντικό, το διάδρομο του Ατλαντικού, διότι ε, όπως είπε και ο συνάδελφος, εγώ είμαι σε ε, μια περιφέρεια που έχει ένα τμήμα αυτού του έργου και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις. Το 2019 μας είπαν στην αρχή, μετά μας είπαν το 2020, ε, στο τέλος και Και τι γίνεται, έχουμε συνεχή κυκλοφοριακή συμφέρουση και παράλυση λόγω των φορτηγών οχημάτων ε, στα σύνορα. Ε, και επομένως τα πάντα τα βρίσκουμε σε μια συνοριακή περιοχή, η οποία είναι απλώ ένα παράδειγμα ε, των όσων συμβαίνουν. Εάν δεν προχωρήσουν αυτά τα προγράμματα, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ούτε στην κοινωνοτομία, ούτε στη βελτίωση του τουρισμού, ούτε στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Η ερώτηση λοιπόν προ του ε, συντονιστέ θα είναι η εξή. Τι μπορούμε να κάνουμε εμεί περισσότερο από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να πετύσουμε από τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν αυτά τα σχέδια προτεραιότητε, διότι πραγματικά μα καθυστερούν πολύ. Ε, θα να ρωτήσω πώ μπορεί να επηρεάσει το έργο του διαδρόμου του ε, ε, μεταξιού το οποίο προχωράει η Κίνα πραγματικά στο σπίτι μας. Εμείς τι κάνουμε, ε, προσπαθούμε να προχωρήσουμε τα σχέδια προτεραιότητας και η Κίνα πραγματικά δημιουργεί το νέο δρόμο του μεταξιού. Ε, και τρίτον, κάτι το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω, και να σας πω μάλλον ότι δεν είναι μόνο θέμα χρηματοδότησης. Πώς μπορούμε να καινοτομήσουμε με ιδιωτική χρηματοδότηση αν μπορούμε να προσδώσουμε ασφάλεια δικαίου σε καμία επιχείρηση και σε κανένα επενδυτή γιατί δεν υπάρχει σαφής τοποθέτηση. Και θα ήθελα να κάνω και μία συγκεκριμένη ερώτηση προς τον κύριο Σέκη για το πώς βλέπει τη στάση της γαλλικής κυβέρνησης, την παρούσα στάση και τις προηγούμενες ε, οι οποίοι δεν θέλουν ε, με κανένα τρόπο να εκτελέσουν το σχέδιο ε, που προβλέπεται μετά από τα σύνορα για να υλοποιηθεί το, ο διάδρομος του Ατλαντικού. Τι μπορούμε να κάνουμε, έχουμε εκθέσεις της Γαλλικής Γερουσίας που από το 2013 και μετά είχε εγκρίνει αυτά τα σχέδια προτεραιότητας και μετά ε, ζήτησε διαφορετικά έργα. Ε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε λοιπόν τη διάθεση, τη θέληση των κρατών μελών. Πρέπει να υπάρξει μια συμμεχία μεταξύ των Ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πιέσουμε τις χώρες να σοβαρευτούν, να χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο αυτούς τους πόρους που είναι ευρωπαϊκοί, αλλά και τους ε, ίδιους πόρους από τον προπολογισμό τους. Κύριε Σέκη, πραγματικά θα ήθελα να μου πείτε τι αξιολόγηση κάνετε εσείς για τις καθυστερήσεις που έχουμε στην Ισπανία από αυτό τον άξονα, τη στάση της γαλλικής κυβέρνησης και επίσης πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σας διότι πραγματικά, συγγνώμη που σας το λέω, ε, είναι λίγο κουραστικό κάθε φορά που γίνεται αναθεώρηση αυτών των έργων να πρέπει να υπενθυμίζουμε τα ίδια πράγματα. Ε, υπάρχουν οι μεγάλοι υπεύθυνοι, τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις ε, κάθε, χρόνο, ε, κάθε χώρας. Ευχαριστώ κυρία Μπελμπάου. Θα μειώσουμε το χρόνο ομιλίας γιατί καθυστερήσαμε πολύ. Γεια σας. Ναι, δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο μας. Εγώ... Έχετε χρόνο, τουλάχιστον τρία λεπτά. Λοιπόν, δεν μου δημιουργείται η αίσθηση μια επίγουσα ανάγκη όσον αφορά το κλίμα από αυτά που έχω ακούσει. Πώ λαμβάνετε υπόψη σα το έργο σα την ανάγκη να απαλλαγούμε πλήρω ε, στι μεταφορέ μα από τον άνθρακα τι επόμενε δεκαετίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη συγκεκριμένη εμπειρία που έχετε αποκομίσει. Ποια είναι τα εμπόδια ε, όσον αφορά την ε, επίτευξη αυτού του στόχου. Εγώ σα δίνω τρία λεπτά και εσεί μιλάτε 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο κύριος Μπέρενσεν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο κύριος Ράιτερς, τα διασυνεριακά έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ολοκλήρωση των διαδρόμων και αυτό είναι κάτι το οποίο ανέδειξαν όλοι οι συντονιστές που μας μίλησαν σήμερα εδώ. Έχουμε και το φάκελο Smart TNT ε, μέσω του οποίου μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε τι διαδικασίε που ακολουθούνται στι επιμέρου χώρε για να αποφεύγονται καθυστερήσει και τα συνεπακόλουθα κόστη. Ε, αυτά βεβαίως ε, όλα εξαρτώνται αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο που δεν φαίνεται να επιταχύνει τις εργασίες του. Θα ήθελα να μου πούν οι συντονιστές πώς αξιολογούν εκείνοι το ντοσχέ αυτό για το δικό τους έργο και πώς ε, πιστεύουν εκείνοι ότι μπορούν να επιταχυνθούν διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτών των διαδρόμων. Και δεύτερον, κύριε Μπάλας, αναφερθήκατε σε 350 έργα. Πόσα από αυτά είναι διασυνοριακά. Ο κύριος Γκρός μας έδωσε κάποια συγκεκριμένα απτά παραδείγματα. Πόσα λοιπόν από τα έργα που αναφέρατε είναι διασυνοριακά και θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα-δυο συγκεκριμένα παραδείγματα όπου πιστεύετε ότι οι διαδικασίες αυτές ε, μεταξύ των διαφόρων χωρών δυσκολεύουν ε, ή διευκολύνουν την ε, επιτάχυνση των έργων. Και Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Τιέν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συντονιστές, πολύ πολύ σύντομα, γιατί η ερώτησή μου έγινε κατά κάποιο τρόπο και από την κυρία Μπιλμπάου και από τον κύριο Ρικέ. Κύριε Σέκη, δείξατε τον χάρτη του διαδρόμου του Ατλαντικού και είπατε ότι το κάτω τμήμα μεταξύ δηλαδή της πόλης του Μπορντό και του συνόρου με την Ισπανία καθυστερεί. Μπορείτε να μας πείτε αν έχετε τρόπο επιτάχυνσης και εμείς σαν κοινοβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε. Όλοι βλέπουμε ότι μεταξύ Μπορντό και Παρισιού η σιδηροδρομική γραμμή υψηλή ταχύτητα έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα πράγματα, κυρίω για τη μεταφορά των ε, επιβατών, αλλά και για τα εμπορεύματα. Βλέπουμε όμως ότι δημιουργούνται νέα σημεία συμφόρηση, όπω λοιπόν είπε και η κυρία Μπιλμπάου, ερωτώ και εγώ τι μπορούμε να κάνουμε για να επιταχύνουμε αυτές τις απαραίτητες υποδομές και διασυνδέσεις κυρίως στις διασυνοριακές περιοχές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τιέν. Εδώ και 30 χρόνια βλέπουμε τι επενδύσεις έχουν γίνει για τις γραμμές υψηλής ταχύτητας. Σήμερα βλέπουμε το τι χρηματοδότηση χρειάζεται. Και αυτό που συνέβη είναι ότι όλα τα κονδύλια επενδύθηκαν στις γραμμές υψηλής ταχύτητας και έχουν παραμεληθεί και εγκαταληφθεί όλες οι υπόλοιπες σιδεροδρομικές γραμμές. Εγώ προτιμώ να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια κονδύλια για την ανακαίνιση κάποιων γραμμών από το να δημιουργούμε διαρκώς νέες γραμμές υψηλής ταχύτητας οι οποίες πραγματικά απορροφούν όλα τα κονδύλια γιατί είναι εξαιρετικά δαπανηρές και σήμερα το ξέρουμε και θα ήθελα να το πω. Η κυρία Αχμό, Καλημέρα σας, έχετε το λόγο. Καλημέρα. Ξεκινάω με μια πολύ σύντομη ερώτηση. Θα παρουσιαστούν και οι άλλοι διάδρομοι. Ή εσείς, κύριοι συντονιστές, μπορείτε να απαντήσετε και για τους άλλους διαδρόμους. Κοιτάξτε, εδώ είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται οι διάδρομοι. Υπάρχουν εννέα, θα υπάρξουν και άλλες ακροάσεις έτσι ώστε να ακούσουμε και τους υπόλοιπους συντονιστές. Πότε θα γίνει αυτό, τις επόμενες ημέρες, με ενδιαφέρει για τις τροπολογίες του 2020. Είμαι μέλος της Επιτροπής προπολογισμού. Πότε, σε ένα μήνα, σε μια εβδομάδα, άμεσα, πότε θα τους ακούσουμε. Είμαι από τη Ρουμανία. Κοιτάξτε, αν δω το χρονοδιάγραμμά μας, δεν έχουμε δυστυχώς συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα. Στην επόμενη συνεδρίασή μας θα προσπαθήσω να έχουμε μια άλλη σειρά συντονιστών για άλλους διαδρόμους. Ναι, αλλά θα είναι πολύ αργά, οπότε θα κάνω τις ρωτήσεις μου τώρα. Εγώ μένω στο Βουκουρέστι. Και όταν έρχομαι στη Γαλλία και στο Βέλγιο, το μισό χρόνο του ταξιδιού μου τον δαπανώ στην εσωτερική μεταφορά για να διασχίσω τη χώρα μου. Δεν συνδέεται η πόλη το Βουκουρέστι με το διευρωπαϊκό δίκτυο. Προσπαθούμε να το πετύχουμε. Εσείς λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει η κατάσταση. Εάν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, η κατάσταση θα είναι η ίδια. Υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες, η Βαλαχία, η Τρανσιλβανία, η Μολδαβία, με 20 εκατομμύρια κατοίκους. Εγώ έχω μια λύση να σας προτείνω και επειδή πραγματικά γνωρίζω την κατάσταση τόπου, χρειάζεται τεχνική βοήθεια. Όταν λέμε τεχνική βοήθεια δεν εννοούμε έγγραφα εννοούμε άτομα τα οποία διαχειρίζονται τα σχέδια. Μέχρι τώρα μας λέγατε πρέπει να αναπτύξουμε τη διοικητική δομή. Αυτό έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα διοικητικά προσόντα, τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό, επαναλαμβάνω, σαν στρατηγική έχει αποτύχει. Και δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο γιατί τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια. Αν συνεχίσουμε με αυτή τη στρατηγική τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να στηρίξουμε την τεχνική βοήθεια με άτομα επιτόπου οι οποίοι μπορεί να είναι Ρουμάνοι αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπάλληλοι της κυβέρνησης της Ρουμανίας, δημόσιοι υπάλληλοι. Ποια είναι η δική σας λοιπόν πρόταση και τι λύση προτείνετε για να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ δυναμική σας ερώτηση. Ο κύριος Κόφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν μια σύντομη προσθήκη στα όσα είπε ο συνάδελφος ε, Κάρινς προηγουμένως. Ήθελα απλώς να ρωτήσω αν γνωρίζουμε σαφώς για τις εκπομπές διοξιδίου του, άνθρακα, ε, του φαινομένου του θερμοκηπίου, συγγνώμη, αυτής της ε, ε, ε κατασκευής. Ε, γιατί έχουμε το κόστος, αλλά δεν έχουμε το κόστος του άνθρακα σε επένδυση σε κεφάλαιο και τις αλλαγές στις εκπομπές που θα οδηγήσουν θα προκύψουν από αυτά τα έργα. Για να έρθω σε συνέχεια με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως, πρέπει να ε, εξαλειφθεί η χρήση του άνθρακα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει πλήρης αξιολόγηση αυτών των έργων, όχι μόνο από οικονομική σκοπιάς, αλλά και από περιβαλλοντικής ε, σκοπιάς ε, και αν έχει υπάρξει μια στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση, μια περιβαλλοντική αξιολόγηση επιπτώσεων. Θα ήθελα μια κάποια απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Κόφ. Ο κύριος Νέβικοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος ως συνήθως. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι συζητιούνται τα ευρωπαϊκά δίκτυα κυρίως ως νέο θέμα της νέας πολιτικής σεζόν και δεν νομίζω ότι υπάρχει και πουθενά καλύτερος χώρος για να πω την άποψή μου. Όσο και πιο ψηφιακό γίνεται ο κόσμος και όσο και αν γίνει περισσότερο ψηφιακό στο μέλλον, πάντα θα χρειαζόμαστε ε, ταχύτερα τρένα, ε, ταχύτερους αυτοκινητοδρόμους, μεγαλύτερους λιμένους, ε, περισσότερα αεροδρόμια, γιατί ζούμε σε ένα πραγματικό κόσμο. Και τα τελευταία χρόνια, πέντε χρόνια στο Κοινοβούλιο, ε, πέρασα πολύ καιρό στην Επιτροπή Προπολογισμών. Παρακολουθούσα τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων και των μεταφορών γενικότερα και διαπιστώνω ότι υπάρχει απλώ έλλειψη χρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε χονδρικά περίπου μισό τρισεκατομμύριο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, συν κάποιες επεκτάσεις ε, πέραν των διαδρόμων και δεν αρκεί η χρηματοδότηση για όλα αυτά. Και ξέρω ότι ο συνολικός ετήσιος προπολογισμός της Ένωσης είναι περίπου 160 ε, δις. Ακόμα και αν δαπανίσουμε λοιπόν όλο τον προπολογισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα δεν θα μπορέσουμε να τα τελειώσουμε γέρος. Και παρεμπιπτόντως, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα είναι σε θέση να ε, χρησιμοποιήσει τόσο μεγάλα ποσά για να ε, καλύψει την υποχρέωση τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων. Και δεν χρειάζεται να αναφέρω εγώ πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη δημιουργία θέσεων εργασία, για την οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν κάποιε χώρε, ιδίω στην περιφέρεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που εξαρτώνται αποκλειστικά από αυτό. Επιχειρήσει που εξαρτώνται από οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Ε, κυβερνήσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσει, δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, ποιοτικό επίπεδο, όλα εξαρτώνται από τι υποδομές. Ε, θυμάμαι μια πολύ δημοφιλή ταινία της δεκαετίας του 90 με τον Ντόμ Κρούζ, ε, στο μεγαλύτερο μέρο τη ταινία φώναζε Show me the money, show the money. Δείξτε μου που είναι τα χρήματα. Αυτό ίσω πρέπει να φωνάξουμε κι εμεί, ε, να υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όλοι εξέφρασαν την άποψή τους Περιμένω λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις για τους στόχους. Δεν χρειάζεται τώρα να συζητάμε χωρίς προσανατολισμό. Χρειαζόμαστε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, ε, ένα ε, καθορισμό για το σχέση με το περιβάλλον, αν έχει υπάρξει αξιολόγηση περιβάλλοντος. Το είπε ο κύριος ε, Ρικέ, ο κύριος Κόφ, ο κύριος Ίσλινγκ για τις συνέπειες για, τον, για το περιβάλλον αλλά και τις κοινωνικές συνέπειες. Τρίτο που είναι σημαντικό και το είπατε όλοι σας, την χρηματοδότηση, την προοπτική χρηματοδότησης ε, που δεν αφορά μόνο το ποσό και ένα μηχανισμό για την απλοποίηση, αν δεν υπάρχουν χρήματα για να προχωρήσουν τα έργα ε, και για να μπορέσετε κι εσείς κάπου να εμπλακείτε, ε, θα γίνουν πολύ σύνθετα τα πράγματα. Και κάτι τελευταίο, και εδώ να μιλήσω στον κύριο Ρόιτερς, διότι έγιναν πολλές ερωτήσεις προς αυτόν, δεν αναφέρθηκε ακριβώς, πάρα πολύ το φλέγον ζήτημα, το θέμα της διαλειτουργικότητας. Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε πλήρη χρήση των δικτύων, όχι όμως σε 10 χρόνια. Ε, πριν από 5 χρόνια ξανασυζητήσαμε το ίδιο θέμα. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε την πραγματική όθηση και να πούμε εδώ στην Κομισιόν Βουδαπέστη-Παρίσι για παράδειγμα. Υπάρχει σύνδεση. Πολύ θα μ' άρεσε. Ε, πώς μπορεί να γίνει λοιπόν αυτό και να μπορέσουμε να πούμε ότι όντως αυτή είναι η Ευρώπη και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λέτε πάντα ότι υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν λόγοι για τη χρηματοδότηση, υπάρχουν λόγοι ε, για το οτιδήποτε. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε όθηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι η αιχμή του δόρατος για να μπορέσουμε να χτίσουμε την Ευρώπη και αυτή την κινητικότητα και αυτή τη διαλειτουργικότητα. Κύριε Ρόιτερς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν το λόγο και χαιρετίζω πραγματικά όλα τα σχόλια που ακούστηκαν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι ε, συγκεκριμένος στις απαντήσεις μου. Πράγματι, έχουμε έναν ξεκάθαρο κανονισμό, ο οποίος εγκρίθηκε στα τέλη του 2013, που λέει ότι αυτό το βασικό δίκτυο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2030 και το συμπληρωματικό έως το 2050 και θα πρέπει να είναι πλήρως διαλειτουργικό η ταχύτητα και ο ρυθμός των επενδύσεων που βλέπουμε και νομίζω ότι είναι ένα σημείο στο οποίο στάθηκαν πάρα πολλοί ευρωβουλευτές, δεν είναι επαρκής. Τα περισσότερα κράτη-μέλη επενδύουν το 0,8% του ΑΕΠ τους, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 1 ή και παραπάνω. 1,2 για την ακρίβεια, του ΑΕΠ του θα έπρεπε να επενδύουν τα κράτη-μέλη για να πετύχουμε του στόχου μα. Οπότε, κύριε Νέβικοφ, που ήσασταν και ο τελευταίο ομιλητή, ναι, είναι σαφή τα πράγματα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερε προσπάθειε για την επίτευξη των στόχων και να ευθυγραμμίσουν τα έργα τους με αυτά που έχουμε διακηρύξει. Αυτό που έχουμε κάνει σε πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή σας είναι να εξασφαλίσουμε επαρκή προπολογισμό. Η συνάδελφός μου Ιάννη ήταν σαφής. Ο προπολογισμό που προτείνεται για το 2020 μπορεί να απορροφηθεί εύκολα. Έχουμε αρκετά έργα τα οποία δεν έχουν χρηματοδοτηθεί καθόλου μέχρι στιγμή, γιατί με τα περιορισμένα μέσα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ιεραρχήσουμε τα πλέον επίγοντα, τα πλέον ευρωπαϊκά αν θέλετε ε, έργα και τα έργα διαλειτουργικότητας, όλα τα άλλα που επίσης είναι απαραίτητα, όπως είναι οι διασυνδέσεις ε, με, την πρωτεύουσα, για παράδειγμα, της Ρουμανίας και όλα αυτά, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μόνο με συνδυασμό προσπαθειών και στο μέτρο του δυνατού. Δηλαδή, ανάμεσα στο ΣΕΦ και το Ταμείο Συνοχής, με το Ταμείο Ιούνκερ, με ιδιωτικά κεφάλαια, έτσι. Αλλά το να έρθω εδώ και να σας πω ε, σήμερα και δεν θέλω να το κάνω γιατί θα υπάρξει ε, σύντομα και μια αναθεώρηση των TNT. Να έρθω εδώ λοιπόν και να σας πω ε, πού βρισκόμαστε. Αυτό ήταν το σημαντικό. Μαζί με τους συντονιστές. Αυτά που μας απασχολούν ιδιαίτερως είναι η διαλειτουργικότητα και έχουμε ορίσει 8 παραμέτρους στο TNT και ο κύριος Γκρότς μας έδειξε πόσο πόσες ελλείψεις υπάρχουν, πόσες αποκλήσεις υπάρχουν, όπως είναι για παράδειγμα και το ίχνος, το εύρος φόρτωσης των ε, τροχών. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε έως το 2030 και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Οπότε θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Πρώτα απ' όλα, το σημαντικότερο είναι να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση. Η νομοθεσία είναι σαφής. Μπορούμε βεβαίω να τη βελτιώσουμε μαζί σας και να την τελειοποιήσουμε σε συνεργασία με εσά. Αλλά αυτό που είναι το σημαντικότερο είναι η χρηματοδότηση. Δεύτερον, προθυμία από την πλευρά των κρατών μελών. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντονιστές μας γιατί προσπαθούν ακριβώς να ε, επιτύχουν ακριβώς αυτό. Έχουμε τις 8 ε, το, τους, τους τις παραμέτρους όπως είπα. Έχουμε τον Brenner η Πατ Κόξ βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που διαχειρίζεται το, το Μπρένερ. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη, είναι και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ο κύριος Πατ Κόξ ε, φέρνει στο ίδιο τραπέζι συζητήσεων το κράτος μέλος, τις εταιρείες, τις κατασκευαστικές, τις ε, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που, μέσα από τις οποίες περνάνε. Αυτά ισχύουν και για τον Μπρένεν, ε, ισχύουν και για όλα τα άλλα έργα. Αν τα κράτη-μέλη δεν δείξουν προθυμία να εργαστούν, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε. Και αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να ρίξουμε λάδι στην ε, μηχανή, προκειμένου τουλάχιστον να ανακοινηθούν τα γρανάζια της, για να μπορέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνεργαστούν μεταξύ τους. Γιατί αν δεν κάνουμε εμείς αυτό, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Και μπορώ να σας δώσω και παραδείγματα για τέτοιων αποτυχιών, αν θέλετε. Τρίτο, Κύριε Ζήλε, σας ευχαριστώ πολύ που ε, αναδείξατε και το, τα βραχυπρόθεσμα ε, αποτελέσματα, αποτελέσματα που πρέπει να, να επιτύχουμε. Ξέρετε, όταν ένας προϋπολογισμός δεν απορροφάται από το κράτος μέλος, τότε αφαιρείται από το κράτος μέλος και δεν ανανεώνεται στον επόμενο κύκλο, στον επόμενο προϋπολογισμό. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να υπάρχουν αναθεωρήσεις και αξιολογήσεις. Αν όμω χρήματα υπάρχουν, έχουν διατεθεί και δεν έχουν απορροφηθεί, τότε αυτά αφαιρούνται. Και αυτή η κατεύθυνση τη Κομισιόν είναι ξεκάθαρη. Το έχουμε ξεκαθαρίσει προ όλε τι κατευθύνσει. ότι εμεί αυτό θέλουμε. Όταν δίνουμε χρήματα, να αξιοποιούνται, να απορροφούνται. Και δεν είναι μόνο το αν ε, ε, ολοκληρώνονται τα έργα στο, στο χρόνο που έχει προβλεφθεί, είναι και το κόστος, είναι και το πόσα χρήματα τελικά έχουν αξιοποιηθεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και τέλος, για την TCT, για τη συνθήκη για τις μεταφορές. Εκεί υπάρχει ήδη μια τεχνική γραμματεία, έχουν γίνει κάποιες πρώτες συναντήσεις μεταξύ των ε, κρατών μελών που συμμετέχουν και ε, ένα από τα, ένα, από τα πρώτα ζητήματα είναι η διασυνορική συνδεσιμότητα. Το Connecting Europe Facility βεβαίως αφορά μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από εκεί για χώρες υπό προσχώρηση, υποψήφιε για ένταξη χώρε κτλ, κτλ. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ακόμη και σε αυτό το επίπεδο να διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά ότι η σημαντικότατη είναι η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η ένταξη συγκεκριμένων έργων στην ολοκλήρωση και στην στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης συγκεκριμένων διαδρόμων. Και σε αυτό πρέπει να γίνουν επενδύσεις όχι μόνο βεβαίως σε ένα συγκεκριμένο τούνελ που θα γίνει στο Μπρένερ αλλά σε ολόκληρο το διάδρομο, σε όλο το μήκος του. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Ρότερς. Ο επόμενος ε, συντονιστής θα πάρει το λόγο σας. Παρακαλώ τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Βλέπετε ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου είναι αποφασισμένα. Θέλουμε αποτελέσματα και θέλουμε και συγκεκριμένη μελέτη αντικτύπου πώς αυτές οι περιοχές που μας αφορούν, από τις οποίες προερχόμαστε, θα συνδεθούν μεταξύ τους. Και η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Τι εμποδίζει σήμερα τη διασύνδεση. Εμείς θέλουμε να ξεκλειδώσουμε αυτά τα σημεία τα οποία σήμερα δυσκολεύουν την πρόσβαση και εμποδίζουν τη διασύνδεση. Το InvestEU αντικατέστησε ένα προηγούμενο πρόγραμμα επενδύσεων στις μεταφορές. Αλλά το θέμα δεν είναι η αντικατάσταση κάτι καινούργιο ή κάτι παλιότερο. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει και πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες. Ξεκινάμε λοιπόν άμεσα με τον κύριο Μπάλας. Κύριε Μπάλας, αλλά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πώς τις διασυνοριακές διασυνδέσεις. Θα σας απαντούσα. Στην κάθε περίπτωση κάνουμε το εξής ερώτημα ποια είναι η προστιθέμενη αξία η ευρωπαϊκή, είτε πρόκειται για μικρό είτε πρόκειται για μεγάλο σχέδιο και πρόγραμμα. Όσον αφορά τώρα την Ιρλανδία και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, όλα αυτά τα διασυνοριακά προγράμματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το ίδιο συμβαίνει εξάλλου και με τον Benelux πρέπει να δούμε και το θαλάσσιο και το ε, κομμάτι των εσωτερικών πλωτών οδών. Και μία άλλη ερώτηση που αφορά τις μακροπρόθεσμες συνεργασίες που έχουμε με τα κράτη-μέλη. Δεν βλέπουμε τις κυβερνήσεις, βλέπουμε τα κράτη-μέλη. Αλλάζει η κυβέρνηση αυτό είναι η δημοκρατία. Υπάρχει μια νέα κυβέρνηση με νέες ιδέες, την οποία βεβαίως κάθε φορά θα πρέπει να πείσουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτές είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεχίσουμε παρακολουθώντας τις αλλαγές. Είπατε κάτι και για την Κίνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της Κίνας. Έχουμε πολύ έντονες συζητήσεις μεταξύ μας, μεταξύ συντονιστών και παρακολουθούμε τις επαφές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών και της Κίνας. Μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει σαν Επιτροπή Μεταφορών το θέμα της Κίνας και της επέκτασης της οικονομικής της επιρροής μέσω των μεταφορών από την γη και από τη θάλασσα. Η Κίνα καλύπτει, αν θέλετε, τις αδυναμίες που έχει στη διασύνδεση και προτείνει πολύ συγκεκριμένες λύσεις με τους γείτονές της, αλλά και με εμάς. Πολύ σύντομα, πιστεύω, μπορείτε να θέσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις με τον νέο επίτροπο. Κανείς δεν ξέρει σήμερα ποιος θα είναι αλλά πιστεύω ότι η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να θίξει αυτό το πολύ περίπλοκο και πολύ λεπτό θέμα που αφορά την Κίνα. Και για λίγο θα απευθυνθώ στον κύριο Ρικέ. Μιλήσατε για τα εργαλεία χρηματοδότησης. Κάνουμε κάθε χρόνο συνεδριάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα των Επενδύσεων και ανταλλάσσουμε εμπειρίες και απόψεις. Έχουμε δύο οικονομολόγους, τον κύριο Σέκη και τον κύριο Μπόντερικ. Οικονομολόγους οι οποίοι έχουν υποβάλει έγγραφα για ε, την εσωτερική συζήτηση αλλά και προς δημοσίευση. Ολοκληρώνω λέγοντας τον κύριο Δίας. Ρωτήσατε πότε μπορούμε να δούμε την υλοποίηση όλων αυτών των σχεδίων. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αν κοιτάξετε το κάθε σχέδιο. Και κάθε φορά βάζουμε τις ημερομηνίες και τα ποσά που αντιστοιχούν. Και λέμε ότι βάσει της αρχής «use it or lose it» ένα κράτος μέλος, εάν δεν μπορέσει να χρησιμοποιήσει, να απορροφήσει ένα συγκεκριμένο ποσό, αυτό χάνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Εγώ θα απαντήσω στην ερώτηση εάν το 2030 θα είχε ολοκληρωθεί αυτή η επένδυση, αυτή η προσπάθεια υλοποίηση των σχεδίων. Η απάντησή μου είναι σαφέστατη. Όχι. Όχι εάν δεν αλλάξουμε μέθοδο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθεί ο διάδρομο εάν η κατάσταση παραμείνει η ίδια στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Α πάρουμε παραδείγματο χάρη το θέμα που αφορά τη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία, Πράγα, Δρέσγη. Η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα μου λένε στην καλύτερη περίπτωση θα έχει ολοκληρωθεί το 2034. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να πιέσουμε τις κυβερνήσεις, τα κράτη. Κάνατε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για του Βουκουρέστη. Εμείς οι συντονιστές τι θεωρούμε το πιο σημαντικό, τη χρηματοδότηση ή τη διαχείριση. Όλοι απαντάμε την διαχείριση αυτών των σχεδίων και δεν μπορούν μόνες τους οι διοικητικές αρχές, οι αρχές της χώρας να υλοποιήσουν. Έχετε δίκιο. Χρειάζονται τα ευρωπαϊκά εργαλεία, χρειάζεται όμως και το καταρτισμένο προσωπικό επιτόπου. Μίλησαμε για την Ελλάδα. Εγώ αν πάρω το δικό μου διάδρομο, οι φάκελοι ΣΕΦ της Ελλάδας χρησιμοποιήθηκαν 100%. Βλέπετε εδώ ότι υπήρχε μια πολύ καλή διαχείριση των προγραμμάτων και μια πολύ αποτελεσματική διαχείριση. Κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει σε όλους τους διαδρόμους, όχι μόνο το δικό μου, πρέπει κάθε φορά όταν βρισκόμαστε σε περιοχές όπως αυτή της Νότιας Ευρώπης να κοιτάμε όλες τις πτυχές της υλοποίησης. Για την Κίνα έχει δίκιο ο συνάδελφος και θα προσθέσω κάτι. Προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι είναι πολιτική ευθύνη των κρατών μελών τα οποία πρέπει κάθε φορά να ξέρουν ποιο οικονομικό εργαλείο θέλουν να αναθέσουν σε κάποιον άλλον. Θέλουν να κρατήσουν τα χαρτιά στα χέρια τους ή θέλουν να τα αναθέσουν σε ξένες δυνάμεις. Και αυτό ισχύει για τα λιμάνια, ισχύει για τους αυτοκινητοδρόμους και βεβαίως το πρόβλημα είναι και η διαχείριση των πόρων, η δημοσιονομική διαχείριση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γνωρίζει τα θέματα αυτά. Για τις μεγάλες επενδύσεις θα πρέπει να εξουδετερώσουμε κάποιες επενδύσεις. Και αυτό είναι μια πολιτική πρόκληση. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και όλα τα κράτη-μέλη να το αντιμετωπίσουν με μεγάλη σοβαρότητα. Αυτό το εύκολο χρήμα που έρχεται από έξω θα πρέπει να χρησιμοποιείται και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς χρησιμοποιείται μου ζητάτε συγκεκριμένες απαντήσεις, σας τις δίνω. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση, κάναμε μία μελέτη με όλες τις χώρες και διαπιστώσαμε ότι θα πρέπει να φτάσουμε τα 486 δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύψει το 1 τρίτο αυτού του τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από τα κράτη-μέλη, από τον ιδιωτικό τομέα και από άλλες πηγές. Η Ευρώπη σας δίνει μία όθηση. Δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τα πάντα. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, σε 25 δις, τα διαρθρωτικά 70 δις για την κινητικότητα και τις μεταφορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας πολύ καλύτερος συντονισμός μπορεί να δώσει μια απάντηση πώς αύριο θα γίνει το Μπρένερ. Πώς θα γίνουν όμως και τα οδικά δίκτυα αυτά που οδηγούν στο Μπρένερ για να απεγκλωβιστούν κάποιες περιοχές. Δεν είναι μόνο αν θέλετε οι μεταφορές. Έχετε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, Δρέσδη Πράγα. Υπάρχει το κομμάτι στην Τσεχία που ουσιαστικά στηρίζεται κατά 80% από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ το γερμανικό τμήμα του έργου αυτού 40% και για τη διασυνοριακή περιοχή αυτή, αλλά και για άλλες όπως ε, την ε, βουλγαρική και ελληνική πλευρά που τους καλούμε σε δύο εβδομάδες ε, στο Ίνσμπρουκ για να συμμετάσχουν στην υλοποίηση αυτού του έργου, του μεγάλου έργου που είναι το Μπρένερ. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν δυνατότητες και δεν πρέπει μόνο να κοιτάμε τις δυσκολίες, αλλά και κάποιες λύσεις, πιθανές λύσεις. Πίεση στα κράτη-μέλη. Ο Χέρελ έδωσε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα αυτό που με ξαφνιάζει πολλές φορές και το λέω ευγενικά είναι ότι το πρόγραμμα εργασιών μας προσυπογράφεται από όλα τα κράτη-μέλη. Όταν περάσουμε όμως την υλοποίηση, εκεί ξαφνικά υπάρχουν κάποιες αδυναμίες υλοποίησης. Κάπως σαν να ξεχνάνε τα κράτη-μέλη τι έχουν υπογράψει. Από τη μία συμφωνούμε όλοι μαζί και μετά διαπιστώνουμε ότι όλα θέλουν να τα αναθέσουν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν συνδράμουν τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ναι, ακούσατε τι είπε ο τελευταίος ομιλητής. Καλό είναι να υπογράφετε, αλλά ακόμα καλύτερο να υλοποιείτε. Φτάνουν οι φλιαρίες. Καλό θα ήταν λοιπόν να συναντόμαστε πιο συχνά έτσι ώστε η Επιτροπή Μεταφορών να μπορεί να κινητοποιήσει κάποια πράγματα. Κύριε Γκρός, κύριε Μπάλας, αυτό το θέμα του δρόμου του μεταξιού είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε πολύ στενά. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα αυτό γιατί υπάρχουν κράτη που προχωρούν με γοργά βήματα και αποφασιστικά βήματα και η Ευρώπη θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσει τουλάχιστον μια ομάδα εργασίας για το θέμα του, των δρόμων του μεταξιού. Κύριε Ρικέ, όπως και με τις επενδύσεις κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ. Θα ολοκληρώσουμε, κύριε Σέκη, μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων, ε, ε, προτάσεις, σχόλια κλπ. Και πάρα πολύ συγκεκριμένε λεπτομέρειες όσον αφορά τους διαφόρους διαδρόμους ε, και τους διαδρόμους που συζητάμε σήμερα. Υπάρχει δυνατότητα, εάν συμφωνεί η Επιτροπή, κατά την παρουσίαση του σχεδίου εργασίας μας, το οποίο θα γίνει σύντομα, ε, μπορούμε να οργανώσουμε κάτι αναδιάδρομο όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Τώρα θα ήθελα να συνεχίσω ε, με μια γενική ερώτηση όσον αφορά τη χρηματοδότηση και κάποιες πιο συγκεκριμένες ε, από εκεί και πέρα. Αυτό που λείπει σίγουρα είναι τα χρήματα. Συμφωνώ με πολλούς για τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που έκαναν. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε εφευρετικοί για νέους τρόπους χρηματοδότησης ε, των ε, έργων μας. Καταρχάς, σε τεχνικό επίπεδο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ε, μόχλευση των διαθέσιμων πόρων, όπως έγινε και με τις προσκλήσεις υποψηφιωτήτων οι οποίες ήταν μικτές ε, και ήταν αρκετά επιτυχείς και ε, φυσικά το ίδιο ισχύει και για τις ε, δυνατότητες blending που ξεκινούν αυτό το μήνα. Επίσης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ποιότητα των προϊόντων θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ και αυτό έχει σχέση και με την ποιότητα των ανθρωπίνων πόρων που είναι διαθέσιμοι για τα θέματα αυτά και πολλά άλλα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα. Χρειαζόμαστε ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ε, καλύτερη ένταξή του στι δραστηριότητές μας και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε και τα κενά. Ε, είναι απαραίτητο να γίνει καλή χρήση των κονδυλίων μας, να αποτελέσουν κίνητρα, αλλά ταυτόχρονα να παρέχουμε και καλά έργα τα οποία είναι κατάλληλα ε, για ε, συνήθεις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Επίσης, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε και καλύτεροι όσο είναι δυνατό σε πρωτοβουλίες σε πιο γενικό επίπεδο. Εδώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα με τη λεγόμενη βιώσιμη ε, πρωτοβουλία χρηματοδότησης. Αυτό ξεκίνησε πέρσι ε, και σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει πολύ σημαντικός αντίκτυπος στις χρηματοδοτικές αγορές. Οι μεταφορές ε, παραβλέφθηκαν, αλλά μετά από επιμονή ε, και καλά επιχειρήματα καταφέραμε πλέον να έχουμε μια κατάλληλη θέση και για τις επενδύσεις που αφορούν τις μεταφορές, οι οποίες φυσικά ε, είναι επιλέξιμες βάσει του γενικότερου τίτλου και να υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πόρων. Αυτές τις εβδομάδες ο νεοεκλογής πρόεδρος ή νεοεκλογής αμαλών πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ξεκινά μια νέα ε, καλή συμφωνία. Ε, τι είναι πιο πολλά υποσχόμενο από τον τομέα των μεταφορών. Ο τομέας των μεταφορών ρηπαίνει μεν πολύ, αλλά ταυτόχρονα μέσω της εξάλληψης της χρήσης άνθρακα στα μέσα μεταφοράς μπορεί να κάνει μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είμαστε κι εμεί όσο το δυνατόν στο προσκήνιο σε αυτέ τι νέε δυνατότητε χρηματοδότηση. Να προσπαθήσουμε επίση να ε, προχωρήσουμε και τα όσα κάνουμε, όπω είπε ο κύριο Ρόιτερ, ε, ε, να παρέχουμε στήριξη, για παράδειγμα, για ηλεκτρικά οχήματα και αντίστοιχε πρωτοβουλίε, καλύτερε ε, μεταφορές ε, ε, επιβατών στον τομέα των αυτιλιακών μεταφορών επίσης να υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG. Κάναμε πολλά στο διαδρομό μου αλλά όχι μόνο σε αυτό και μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη. Και επίσης κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θίξατε. Ένα αφορά την Ισπανία και τη Γαλλία. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος για το πολύ ε, κρίσιμο πρόβλημα το οποίο έχει σχέση με τη γαλλική απόφαση να αναβληθούν πάρα πολλά έργα ε, μπορέσουμε να συστήσουμε μια υψηλή επίπεδου διπουργική ομάδα η οποία ε, συναντιέται τακτικά ε, η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου για να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τη μεταβατική περίοδο και κυρίως ε, για την αναβάθμιση ε, το τμήματος Bordeaux ε, και το τμήμα των συνόρων του Ντάξ και φυσικά ε, υπάρχει και μία πρόταση για, αυτο, για σιδηρόδρομο από τη Βικτόρια στη Λίλ πρέπει να αναβαθμιστεί η παρούσα γραμμή και επίσης έχουμε κατά νου το γεγονός ότι πρέπει να συνδέσουμε Ανατολή-Δύση, όχι μόνο Δύση-Βορανότο. Και ε, επιμένουμε, όπως είπε και ο κύριος Ρόιτερς, ότι οι δύο χώρες ε, θα πρέπει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο να συζητούν και να βρουν κατάλληλες λύσεις. Το αυτό ισχύει βεβαίως και μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας. Ε, το 2030 απέχει πολύ μεν, αλλά πρέπει να επιμείνουμε ότι όσα το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος γίνει, ε, είναι πολύ σημαντική, διότι χάθηκε χρόνος ε, με την κρίση κυρίως στην Πορτογαλία και πρέπει κάπως ε, να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο. Δεν πρέπει να ανακόψουμε την πρόοδο και νομίζω ότι μπορώ να σας πω και ίσως ε, αν μπορέσουμε να συναντηθούμε και για το πρόγραμμα εργασία, θα έχω περισσότερο χρόνο και θα μπορέσω να είμαι πιο συγκεκριμένο. Αλλά υπάρχει κάποια πρόοδο. πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε, να καταλάβουμε για ποιου λόγου υπάρχει καθυστέρηση. Ε, δεν είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν καθυστερήσει, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο να μην γίνεται τίποτα. Ε, και κάποια προσωρινή λύση, ε, εν αναμονή της οριστικής λύσης, ε, είναι σίγουρα καλύτερη από το τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σέκη. Νομίζω ότι μπορούμε να χειροκροτήσουμε τον κύριο Ρόιτερς και τους τρεις συντονιστές, ε, τους κύριους Γκρός, Μπαλάς και Σέκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Το συμπέρασμα είναι ότι εμάς περιμένει πολλή δουλειά. Ε, με πολύ συντονισμένο τρόπο και κυρίως ε, στα τεχνικά ε, θέματα, στα θέματα προϋπολογισμού, αλλά επίσης δεν συζητήσαμε και πάρα πολύ τα υπόλοιπα, την ψηφιοποίηση, την εξάλληψη της χρήσης άνθρακα. Υπάρχουν και όλα αυτά τα θέματα της διαλειτουργικότητας, το είπα, διότι δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων και επομένως πρέπει να γίνουν κάποια παραπάνω, ώστε οι διάδρομοι αυτοί πραγματικά να μας δώσουν μία οδό, δεν κάνουμε πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρκετά κατά την άποψή μου, και να προσπαθήσουμε να συνεργαζόμαστε και με τα κράτη-μέλη. Σίγουρα μπορείτε να βασιστείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βεβαίω. Σα ευχαριστούμε για την παρουσία σα και η πάρτα τη Ευρωπαϊκής Επιτρο... της Επιτροπή μα θα είναι πάντα ανοιχτή εδώ και ελπίζω να σα δω σύντομα. Σα ευχαριστώ πολύ. Allez, nous Συνεχίζουμε λοιπόν και θα ζητήσω τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, τον κύριο Μπάουερ, να έρθει στο βήμα. Κύριε Φέρμπερ, καλημέρα. Allez, nous continuons, s'il vous plaît. Συνεχίζουμε. Μπορείτε να βγείτε εάν θέλετε να συνεχίσετε τις συζητήσεις σας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι αυτό που αφορά την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Ήρα, με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Διευθυντή Τζόζεφ Ντόπελμπάουερ. Ο ρόλος σας είναι διπλός. Έχετε ένα τεχνικό ρόλο με το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, με το οποίο έχουμε εισάγει νέες αρμοδιότητες και αποστολές, όπως οι άδειες, το θέμα των εξοπλισμών, η διαχείριση της κυκλοφορίας, το ERTMS που είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών, η επέκταση των αρμοδιοτήτων τας βεβαίως έχουν, έχει μεγάλες συνέπειες και όσον αφορά τους εξοπλισμούς και το προσωπικό. Και φυσικά το δημοσιονομικό τμήμα μπορείτε να μας παρουσιάσετε την υλοποίηση των προγραμμάτων, τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε, γιατί όπως ξέρετε εδώ στην Επιτροπή μας στηρίζουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τις οποίες θεωρούμε ύψιστη προτεραιότητα. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Κατόπιν, κύριε Ντόπελμπάουερ, μπορείτε να απαντήσετε πολύ συγκεκριμένα στις ερωτήσεις που θα σας απευθύνουν τα μέλη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και έχω τη δυνατότητα να σας εξηγήσω την κατάσταση στην οποία που βρισκόμαστε, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαϊκός Σιδηρόδρομος. Θα σας εξηγήσω επίσης τη σημασία που έχουν οι σιδηρόδρομοι για ένα πιο πράσινο σύστημα μεταφορών καθώς και τη συμβολή ε, που μπορεί να ε, συνεισφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο δεν είμαι σε θέση να σας εξηγήσω στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτούς θα σας πρότεινα να ε, τους ρωτήσετε, να, τις σχετικές ερωτήσεις να τις θέσετε στον ε, υποψήφιο επίτροπο που θα αναλάβει το σχετικό φάκελο. Πολύ σύντομα λοιπόν, η κατάσταση του σιδηροδρόμου είναι η εξή. Υπάρχουν πλεονεκτήματα, υπάρχουν και μειονεκτήματα. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, θέλω να τονίσω ιδίω δύο στοιχεία. Πρώτον, είναι η πολύ υψηλή ασφάλεια. Αν, αν συγκρίνεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου με τις οδικές μεταφορές, υπάρχει ένα επίπεδο ασφάλειας που είναι 50 φορές πάνω από, για το σιδηροδρόμο από ό,τι, ε, από ότι οι οδικές ε, μεταφορές. Το άλλο στοιχείο είναι η εξάλληψη του άνθρακα. Εδώ το πλεονέκτημα των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερο έναντι των οδικών μεταφορών και των αερομεταφορών. Ωστόσο, αυτά τα πλεονεκτήματα συνοδεύονται και από δύο βασικά μειονεκτήματα. Πρώτον, είναι ο ανταγωνισμός που δέχεται ο σιδηρόδρομος από άλλους τρόπους μεταφορών και αυτός είναι ένας ανταγωνισμός που βασίζεται σε μια ε, μη ισορροπημένη κατάσταση αν θέλετε και δεύτερον και αυτό είναι και ο, ο βασικότερος τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός μας είναι ο καταρκερματισμός του Ευρωπαϊκού Συνδρομικού Συστήματος. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον Άκουσα λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση που έγινε γύρω από τους διαδρόμους. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη της Ευρώπης με όλους τους συνοριακούς σταθμούς στο σιδηρόδρομο. Και ξέρετε ότι ο προκάτοχος της κυρίας Ντέλη, ο κύριος Κράμερ, είχε θέσει στόχο του να κλείσουμε αυτά τα κενά που υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πάρα, ε, σημεία συνοριακής διέλευσης στο σιδηρόδρομο που ε, είτε λείπουν είτε δεν υπάρχουν πια. Ένα από αυτό είναι και η σιδηροδρομική σύνδεση του Βαλενσιάν, που είναι και, όπου είναι και η έδρα του οργανισμού μας με τις Βρυξέλλες. Υπήρχε αλλά δεν υπάρχει πια. Επίσης, άλλο πρόβλημα είναι ότι αν υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση, δεν υπάρχει ένα συνεκτικό σύστημα τεχνικών και λειτουργικών κανόνων. Μιλώ για την διαβόητη διαλειτουργικότητα την οποία ανέφερε και η κυρία Πρόεδρος εδώ στην προηγούμενη συζήτηση. Και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι ο σιδηρόδρομος είναι ο μόνος τρόπος μεταφορών, το μόνο είδος μεταφορών για το οποίο δεν υπάρχουν γενικοί παγκόσμιοι κανόνες. Στα φορτηγά, για παράδειγμα, άμα θέλει να μεταφέρει εμπορεύματα από την Ουκρανία μέχρι την Πορτογαλία, το φορτηγό μπορεί να διασχίσει την ε, διαδρομή αυτήν χωρίς ε, τεχνικά ή λειτουργικά εμπόδια. Αν θέλετε όμως να πάτε τρένο από την Ουκρανία στην Πορτογαλία, τότε θα σταματήσετε ήδη στα πρώτα σύνορα με την, με την Πολωνία, γιατί το άνοιγμα των τροχών είναι διαφορετικό. Ο βασικός τομέας λοιπόν στον οποίο έχει δραστηριοποιηθεί ο οργανισμός μας είναι η επίλυση των προβλημάτων που εμφανίζονται στα σύνορα. Και εδώ έχω παραθέσει έναν αριθμό ζητημάτων που βρίσκει κανείς σε όλα τα σημεία διασυνοριακής διέλευσης και αφορούν όλους τους διαδρόμους. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες, υπάρχουν διαφορετικές δοκιμές, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικά συστήματα εποπτείας. Και όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει επιτακτικά να ε, επιληθούν αν θέλουμε να εξαλείψουμε από τις μεταφορές τον άνθρακα. Οι μεγάλες αποστάσεις εξορισμού περιλαμβάνουν διασυνοριακές διελεύσεις. Για τις μικρότερες αποστάσεις δεν υπάρχει λόγος πια να χρησιμοποιούμε αεροπλάνα. Θα μπορούσαμε να ε, μεταβούμε όλοι στο σιδηρόδρομο. 800 χιλιόμετρα μπορεί εύκολα κανείς να τα, διανύσει μέσα σε 4 ώρες. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να επιληθούν αυτά τα διασυνορικά προβλήματα που υπάρχουν. Και εδώ ακριβώ έρχεται να δραστηριοποιηθεί ο οργανισμό μα. Δραστηριοποιούμαστε με άλλα λόγια στον τομέα των... τη τεχνική και λειτουργική επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να τυποποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σιδηροδρόμων και να του δώσουμε το χαρακτήρα ενός ενιαίου χώρου σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, ο οργανισμός μας ιδρύθηκε το 2004. Υπάρχουμε λοιπόν εδώ και 15 χρόνια. Έχουμε 170 μέλη στο προσωπικό μας. Έδρα μας είναι το Βαλενσιάν στην Γαλλία. Έχουμε ε, εγκαταστάσεις συνεδριάσεων στη ΛΥΛ. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε πιο ελκυστικό και πιο βιώσιμο τον σιδηρόδρομο για την κοινωνία και έχουμε πρόσφατα διευρύνει την εντολή μας με σκοπό να γίνουμε Ευρωπαϊκή Αρχή. Με το, με το τέταρτο πυλώνα του πακέτου για την ε, κινητικότητα. Από τις 16 Ιουνίου 2019 ο οργανισμός μας έχει πλέον ε, ευθύνη να εκδίδει εγκρίσεις τύπου που έχουν ισχύ σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι, ευρωπαϊ... είναι ιστορική κοινοτομία. Θυμηθείτε το χάρτη που σας έδειξα πριν με τα σύνορα. Είναι η πιο σημαντική αλλαγή στη σιδηροδρομική νομοθεσία που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Για πρώτη φορά έχουμε πλέον μια ευρωπαϊκή αρχή η οποία μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά και εγκρίσεις που, είναι, ε, που έχουν ισχύ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πορεία της περαιτέρω εναρμόνισης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Σιδηροδρόμων. Τώρα, η κατάσταση είναι εξή. Από τα 28 κράτη-μέλη, δύο δεν εμπίπτουν στο πεδίο ε, εφαρμογή των δικών μας δραστηριοτήτων, γιατί η Μάλτα και η Κύπρος δεν έχουν σιδηρόδρομο. Μόλις τα 8 κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει έως τις 16 Ιουνίου την, ε, τις οδηγίες για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα. 18 κράτη-μέλη ζήτησαν μια μονοετή παράταση και θα μεταφέρουν τις συγκεκριμένες οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 16 Ιουνίου του 2020. Πρέπει να πω ότι για τον οργανισμό μας αυτό ήταν, μια... ήταν κακή και καλή είδηση ταυτόχρονα. Κακή είδηση διότι προφανώς ε, πρόκειται για καθυστέρηση της διαδικασίας, περιπλέκει ε, τα πράγματα, γιατί για κάποιες χώρες και για κάποιους διαδρόμους υπάρχουν ταυτόχρονα δύο νομικά καθεστώτα υπό τα οποία εμπίπτουν. Είναι όμως και κακή είδηση για τη χρηματοδότησή μας. Γιατί εμείς καλούμαστε να καλύψουμε μέρος των ε, δραστηριοτήτων μας των δραστηριοτήτων που σας έλεγα για την πιστοποίηση και την έγκριση και να καλύψουμε μόνοι μας τα, το κόστος που, χρησιμο, που προκαλείται. Ε, όταν μόλις 8 κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει στο Εθνικό του Δίκαιο την οδηγία, καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν επαρκούν. Η θετική πλευρά από την άλλη μεριά είναι ότι μόλις με 8 κράτη-μέλη είχαμε μια ομαλή έναρξη αν θέλετε. Είχαμε τόσα όσα έργα χρειαζόταν να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, εκείνα τα χρήματα που ακριβώς μας επαρκούσαν για να ξεκινήσουμε αν θέλετε τη δουλειά. Από τον Ιούνιο του 2019 όλα τα βαγόνια, τα εμπορευματικά πρέπει να περνάνε από τον οργανισμό μας σε αυτά τα 8 κράτη-μέλη που σας είπα και που εμφανίζονται εδώ με πράσινο. Σημαντικό στοιχείο, και μπορείτε να το, να το έχετε ακούσει ήδη ως όρο, είναι αυτό το one-stop shop, η ενιαία θηρίδα. Ένα σύστημα ενημέρωσης και επικοινωνίας που είναι πλέον το μοναδικό σημείο πρόσβασης για όλες τις εγκρίσεις και όλες τις πιστοποιήσεις που δίνονται στην Ευρώπη. Ανεξάρτητα από το αν η αρχή, ο οργανισμός μας είναι αυτός που εκδίδει την έγκριση την πιστοποίηση ή αν είναι κάποια εθνική αρχή. Όλες οι αιτήσει πρέπει να περνάνε μέσα από αυτό το One Stop Shop που είναι ένα εργαλείο, ένας μηχανισμός που τον ανέπτυξε και τον ε, συντηρεί ο οργανισμός μας. Ήταν μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο μερικώς και πλέον βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τις 16 Ιουνίου. Η τρέχουσα διαθεσιμότητα του εργαλείου αυτού είναι 98,7%. Από τις 16 Ιουνίου λοιπόν φέτος είχαμε μόλις 7 ώρες μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και αυτά, αυτές οι ώρες ε, οφείλονταν ε, σε προβλήματα που ε, αν, αντιμετώπισε ε, ο ε, φορές που είχε αναλάβει την έκδοση των εγκρίσεων. Στόχος μας είναι 99% διαθεσιμότητα. Έχουμε λάβει ε, 100 αιτήματα ε, έως την Παρασκευή. Έχουμε εγκρίνει 92 και λάβαμε την τελευταία Παρασκευή και τα πρώτα χρήματά μας. Τα πρώτα 9.000 ευρώ λάβαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Λοιπόν, θα παρακάμψω κάποιες από τις ε, διαφάνειες που είχα ετοιμάσει για να μην σπαταλήσω το χρόνο και θα περάσω κατευθείαν στις προκλήσεις που έχω προετοιμάσει να σας παρουσιάσω. Δεν θα σας μιλήσω για το ERTMS. Το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αφορά τον προϋπολογισμό και τους πόρους μας. Εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ένα δομικό πρόβλημα, διαρθρωτικό, γενικό, και το άλλο αφορά την έναρξη των εργασιών μας. Το δομικό, το διαρθρωτικό πρόβλημα ήταν το γεγονός ότι Μα ανατέθηκαν περισσότερα καθήκοντα από ό,τι μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα από αυτά ήταν και το One Stop Shop, το οποίο αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2016, αλλά δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη ε, στον προϋπολογισμό της Κομισιόν. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να καλύψουμε από ίδιους πόρους μας 1,2 εκατομμυρίων ευρώ ε, το κόστος για τη δημιουργία και τη συντήρηση αυτού του μηχανισμού. Αυτό σήμαινε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούσαμε να καλέσουμε εμπειρογνώμονες... για να... στις συνεδριάσεις μας. Δεύτερο, στη φάση έναρξης έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε τιμολόγια μόλις αφότου ολοκληρώσουμε το κάθε έργο και από εκεί και πέρα πρέπει να πληρωθούμε εντός 60 ε, ημερών. Δηλαδή για τα έργα που ξεκινάνε την 1η Ιανουαρίου του 2019, τα πρώτα χρήματα τα λάβαμε μετά το ε, τέλος του Φεβρουαρίου. Αυτό είναι ένα θέμα, θέμα ροής ε, ταμιακής που ε, θα μας δημιουργήσει προβλήματα και στο μέλλον, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ε, τη βεβαιότητα ότι πάντοτε θα υπάρχει μια σταθερή ροή ε, έργων και αιτήσεων. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να δημιουργηθεί ένα μαξιλαράκι, ένα αποθεματικό αν θέλετε, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πάντοτε θα μπορούμε να καλύπτουμε το κόστος και τα έξοδά μας. Με αυτό το νέο καθεστώς του οργανισμού λοιπόν, πραγματικά μπήκαμε σε μια νέα εποχή σε μια νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο. Συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου σιδηροδρόμων. Έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι με αυτή την ενιαία ευρωπαϊκή αρχή πιστοποίησης και έγκρισης δίνουμε όθηση στην τάση εναρμόνισης και τυποποίησης γιατί εμείς πάντοτε θα αποφασίζουμε στη βάση των ευρωπαϊκών κανονισμών και κανόνων και όχι στη βάση εθνικών κανονισμών και κανόνων. Και επί αυτής της βάσης μπορούμε να θέσουμε τα θεμέλια για μια αποτελεσματική απαλλαγή από τον άνθρακα στις ευρωπαϊκές μεταφορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Euh, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή, αλλά και για, κυρίως για την επαγρύπνηση την οποία μας καλείτε να λάβουμε υπόψη. Θέλουμε να στηρίξουμε τους σιδηροδρόμους στην Ευρώπη. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Και δίνω το λόγο αμέσως στον κύριο Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ερωτήσεις. Πόσους διαδρόμους για μεταφορές εμπαρευμάτων Πρόκειται να αναπτύξετε. Επίσης, με αυτό το one-stop shop θα προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδρομές και οι μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών από την Ελλάδα μέχρι τη Βόρεια Γερμανία. Τι έχετε να πείτε για τη διαλειτουργικότητα και ποια είναι η συνολική σας στρατηγική Μιλάτε για διαλειτουργικότητα. Πώς θα είναι η κατάσταση σε 5, 10, 15 χρόνια, σύμφωνα με εσάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαριουνέσκου. Ο κύριος Ραμόντιας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Ντόπελ για την παρέμβασή του, γιατί νομίζω ότι ήταν μια ε, παρέμβαση η οποία διευκρίνησε πάρα πολλά πράγματα. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο σιδηροδρομικό τομέα εξακολουθεί να είναι ένα τομέα πολύ μεγάλη οικονομική σημασία, διότι επιτρέπει ε, κοινωνική και εδαφική συνοχή, αλλά όπω βλέπουμε ε, και ένας τρόπος για να δράσουμε ε, και να αντιμετωπίσουμε, να μετριάσουμε τις ε, περιβαλλοντικές και κλιματικές αλλαγές. Ε, η Ισπανία έχει τρένο υψηλής ταχύτητας. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να σας εκφράσω ως ανησυχία της ομάδας μου είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν τηρούν τα θέματα της εφαρμογής των σιδηροδρομικών πακέτων. Ε, το γεγονός ότι δεν τηρούνται και δεν έχουν συμπληρωθεί σημαίνει ότι θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Για τους ε, φιλελευθέρους επίσης ε, ε, τίθεται και θέμα του ελεύθερου ανταγωνισμού και η σταδιακή απελευθέρωση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Και το πιο σημαντικό είναι το γεγονό ότι δημιουργούνται ατυχήματα και τα ατυχήματα ορισμένε φορέ είναι και θανατηφόρα. Και το Renew Europe και οι Ciudadanos, στους οποίους ανήκω, ε, ε, θα ήθελε να εκφράσει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων ε, ενός ατυχήματος που έγινε στην Ισπανία, του τρένου στη Γαλλικία το 2000 13 ε, είχαμε 30 νεκρούς και 114 ε, στραυματίες Και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτό το συγκεκριμένο ατύχημα, ε, κύριε Ντόπερ Μπάουερ, διότι βλέπουμε πώς οι χώρες μέλη και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν έλαβε υπόψη τα αιτήματα για ανεξάρτητες τεχνικές έρευνες, τεχνικές έρευνες που ζήτησε και ο οργανισμός σας. Όσον αφορά αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο γεγονό ε, και αυτό στο οποίο αναφερθήκατε εσεί ε, για την εναρμόνιση του σιδηροδρομικού κλάδου, θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Τι μέτρα σκοπεύετε να ε, εφαρμόσετε ή τι μέτρα σκοπεύει να έχει ο οργανισμό σα για να μην υπάρχει μη τήρηση των κανονισμών. Γιατί αυτό το γεγονό ότι δεν τηρούνται οι κανονισμοί είναι κάτι το οποίο αποτρέπει το βασικό ε, στοιχείο για το οποίο δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ραμόν Δίαθ. Ε, ε μια ενημέρωση για τους καινούριου. Εάν τα κράτη-μέλη τα 18 δεν εφαρμόζουν την τρίτη δέσμη ε, μέτρων για τους σιδηροδρόμους μέχρι το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει διαδικασίε επί παραβάση. Θα πρέπει λοιπόν κάπως να κινηθούν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ξεκινάει αυτές τις διαδικασίες επί πολύ συχνά ε, μπορεί να ε, και πολύ ακριβά στα κράτη-μέλη. Ο κύριος... Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας από πλευράς Πρασίνων και Ευρωπαϊκής ε, Ελεύθερης Συμμαχίας. Ε, χαιρετίζουμε την προσέγγισή σας ε, για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών γραμμών στην Ευρώπη και εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα ε, με τα στοιχεία ασφαλείας που μας δώσετε για τους σιδηροδρόμους και κυρίως για την περιβαλλοντική συμβολή της μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μέσω σιδηροδρόμων. Και καλωσορίζουμε το γεγονό ότι η τυποποίηση είναι πρώτων πυλών, αλλά βέβαια ανησυχούμε για αυτά τα 18 κράτη-μέλη. Το ερώτημα είναι κατά πόσον είστε αισιόδοξο ότι τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν αυτά τα νέα πρότυπα μέσα σε ένα χρόνο ίσως ή σε 12 με 18 μήνες. Είστε αισιόδοξο ότι όντως θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και μια δεύτερη ερώτηση. Έχετε κάποιες σκέψεις ε, ή σας ανησυχεί το θέμα της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Έχει άποψη ο οργανισμός σας ε, και για τον αντίκτυπο ε, που έχει αυτό στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσίαση. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας για τη βελτίωση των σιδηροδρόμων στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ο κύριο Καμπομενώση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα Ιταλικά. Η Ιταλία και η Γαλλία, όπως είδαμε, είναι μεταξύ των λίγων χωρών που μετέφεραν την οδηγία για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα ε, και μάλιστα αρκετά σύντομα. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πού βρισκόμαστε όσον αφορά την έγκριση χρήσης ε, τρένων μεταξύ των δύο χωρών, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς ενός ε, Ιταλού ε, παρόχου. Το Μιλάνο και το Παρίσι είναι δύο πόλεις οι οποίες χρειάζονται μιας κάποιας μορφής σύνδεση και για εμπορικούς λόγους, αλλά και για άλλους οικονομικούς λόγους και πιθανόν διάδρομος ε, το Ρήνο Λιόν που θα επιταχύνει περισσότερο τις διαδικασίες. Πρόκειται όμως για κάτι το οποίο θα μπορούσε ίσως να λειτουργεί ε, το 2020 και θα μπορούσε να βοηθήσει αυτές τις δύο πόλεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Κύριε. Σας ευχαριστώ κύριε Ντόπελμπαουρ για την παρουσίασή σα. Εγώ είχα την τιμή πριν από δύο χρόνια να είμαι ο εισηγητής ε, για τα ρυθμιστικά και κανονιστικά θέματα που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Μπορείτε να μας πείτε όσον αφορά τα θέματα της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας υπάρχει καθυστέρηση, αλλά δεν νομίζω ότι <laughs> αν συγκρίνουμε την κατάσταση με αυτό που συμβαίνει σε άλλους τομείς υπάρχει εδώ θέμα για κυρώσεις. Όσον αφορά την εναρμόνιση χιλιάδων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν ε, τις διαφορετικές χώρες και το εθνικό επίπεδο. Πώς εξελίσσεται αυτό το έργο. Και βεβαίως εδώ σίγουρα χρειάζεται και επιπλέον προσωπικό και επιπλέον χρηματοδότηση. Για το 2020 είπατε ότι προχωράει το θέμα της μεταφοράς των εμπορευμάτων. Όμως, στην βάση δεδομένων σας δεν υπήρχε απολύτως τίποτα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα βαγόνια που αφορούν τη μεταφορά των εμπορευμάτων και τις προδιαγραφές τους 1435 ή 1535. 15-20 τελικά ποια είναι η επιλογή σας όσον αφορά τις τεχνικές αυτές προδιαγραφές. Κύριε Πίπερ, είστε στο τηλέφωνο ή θα μιλήσετε. Έχετε το λόγο. Όχι, μην ανησυχείτε κυρία Πρόεδρε. Εγώ πάντα σας ακούω. Το θέμα τώρα του οργανισμού σιδηροδρόμων. Έχετε και άλλες δυσκολίες. Σκέφτομαι από τη στιγμή που τα χρήματα της πιστοποίησης έχουν δοθεί. Βλέπουμε σήμερα μόνο 8 κράτη-μέλη να έχουν μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία και βλέπουμε ότι πάρα πολλές χώρες, τις οποίες δεν θα κατανομάσουμε, ε, δεν έχουν καθόλου προχωρήσει όσον αφορά τη μεταφορά. Όσον αφορά τις διαδικασίες η παραβάση, υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν τέτοιες προσφυγές. Εγώ παρακολουθώ το θέμα αυτό εδώ και 10 χρόνια και έχουμε αρχίσει λιγάκι να ανυπομονούμε. Νομίζω ότι έχει παρατραβήξει λίγο αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πίπερ. Ο κύριος Στερικέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετώ τον ε, Ζώσεφ Ντόπελμπάουρ και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που ίσως φανεί λεπτομέρεια και έχει άμεση σχέση με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Ο κύριος Διευθυντής ε, του οργανισμού αναφέρει ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Αυτό είναι πραγματικά εξωφρενικό. Το 2004 αυτός ο οργανισμός που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια δεν συνδέεται ακόμα με τις Βρυξέλλες. Δηλαδή, η πόλη της Βαλοσχέν και οι Βρυξέλλες έχουν ακόμη προβλήματα άμεσης διασύνδεσης. Υπάρχουν 7 χιλιόμετρα τα οποία ακόμα δεν καλύπτονται. Κύριε Ντόπελμπάουερ, σας κάνω λοιπόν την ερώτηση πόσο προσωπικό επιπλέον θα χρειαστείτε τη στιγμή που θα αρχίσει η επεξεργασία του τετάρτου πακέτου για τους σιδηροδρόμους. Δεύτερη ερώτηση. Έχετε κάποια νέα από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις προσλήψεις καθώς και την περιορισμένη διάρκεια και περιορισμένο αριθμό των συμβάσεων, γιατί βεβαίως οι συνεργάτες με προσόντα τα οποία θα θέλατε, τους οποίους θα θέλατε να προσελκύσετε και να προσλάβετε, πολλές φορές διστάζουν να δεχτούν μία σύμβαση ορισμένου χρόνου, περιορισμένου θα έλεγα χρόνου, που μπορείτε σήμερα να τους προσφέρετε. Ο κύριος Ντέλη. Ένα σύντομο ερώτημα. Μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους αυτά τα κράτη-μέλη, τα 18, ζήτησαν παράταση της προθεσμίας που είχαν για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Και ποιο ήταν το πρόβλημα στον υλικό εξοπλισμό. Προφανώς τα εμπορεύματα ήταν πρόβλημα, αλλά ίσως υπήρχαν και άλλα ζητήματα στον υλικό εξοπλισμό που δημιούργησαν προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη. Είπατε και στις διαφάνειες ότι έχετε 170 εργαζόμενους προσωπικό. Πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους συνεργάζονται με τα 8 αυτά κράτη-μέλη με τα οποία συνεργάζεστε ήδη, πόσο περισσότερο προσωπικό θα, θα χρειαστείτε από του χρόνου, αν όλα πάνε καλά βεβαίω. Κύριε Ταλέρ, ευχαριστώ. Κύριε Ντόπλεπα, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι εδώ σε αυτή την αίθουσα όλοι ευχόμαστε ο σιδηρόδρομος να γίνει ακόμα πιο επιτυχημένος, να μπορέσει να ε, διατηρήσει την λειτουργία του, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο καθιστώντας πιο ακριβές τις οδικές μεταφορές. Αντιθέτως, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα των σιδηροδρόμων και επενδύσεις. Και εσείς ο ίδιος ε, άλλωστε ε, αναφέρατε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Ε, ο σιδηρόδρομος. Θα με ενδιέφερε ε, να μου πείτε ε, τι, τι χρήματα θα χρειαστούν για να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στα σημεία συνοριακής διέλευσης. Είτε αφορά το ίχνος, το άνοιγμα των τροχών, είτε αφορά τις, τα γλωσσικά ζητήματα πώς μπορούμε να ε, ξεπεράσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια προστατευτισμού, πώς μπορούμε συνολικά να οφειλήσουμε την, τον σιδηρόδρομο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάλερ. Μην ξεχνάτε ότι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του σιδηροδρόμου είναι οι αεροπορικές μεταφορές με εντελώς διαφορετικά βάρη. Ας πούμε λοιπόν τα πράγματα ως έχουν. Πρόκειται για αθέμητο ανταγωνισμό από μέρους των αεροπορικών μεταφορών που σήμερα βλέπουμε να απορροφά εξαιρετικά πολλά κονδύλια τα οποία δεν κατανέμονται όπως θα έπρεπε στους σιδηροδρόμους. Ο κύριος Νιούτον δεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είπατε α, για αυτό το τρένο που πηγαίνει από την Ουκρανία στην Πορτογαλία στην ε, Πολωνία, συγγνώμη, όπου υπάρχει διαφορά στο άνοιγμα τροχών. Υπάρχει ελπίδα τα επόμενα 20 χρόνια να υπάρχει ενιαίο άνοιγμα τροχών, γιατί υπάρχει και άλλο άνοιγμα για, για, τους, για τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Ποιο είναι το όραμα που μπορείτε να μας δώσετε εσείς. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κυρία Μπιλμπάου, έχει το λόγο. Ναι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξηγήσεις σας. Και νιώθω και ευγνωμοσύνη και λίγο απεσιοδοξία, γιατί εγώ ήμουν εισηγήτρια της έκθεσης για τη διαλειτουργικότητα και θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη συνεργασία που είχαμε, πάνω από δύο χρόνια δουλειάς και πολύ ενδιαφέρον για να ξεκινήσει ένα πακέτο από πολιτική σκοπιά ε, και τελικά καταφέραμε να διατηρήσουμε και χάρη σε αυτό έχουμε την ενία θηρίδα και μια σειρά από διαδικασίες οι οποίες ξεκίνησαν. Η ερώτηση μου είναι η εξή. Οχτώ χώρε έχουν εφαρμόσει του κανόνε για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα. Οι 18 υπόλοιπε πιστεύετε ότι εργάζονται για την εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία και χρειάζονται χρόνο, ή πιστεύετε ότι πρόκειται για μία ακόμα πρακτική προστατευτισμού η οποία θα μπορούσε και να παραταθεί. Ε, ζήτησαν συνεργασία από τον οργανισμό για να εφαρμόσουν ε, σωστά την νομοθεσία. Δεύτερον, ε, ακούσαμε πάνω από 11.000 διαφορετικούς κανόνες οι οποίοι είναι διάσπαρτοι ε, μεταξύ των κρατών μελών. Ο στόχος ήταν να υπάρξει εναρμόνιση και να μειωθούν οι κανονισμοί, να είναι 200 ή 300 οι κανόνες. Ε, πώς ε, προχώρησε η δουλειά, υπήρξε όντως η μείωση, μέχρι ποιου σημείου επιτεύχθη ο στόχος. Και επίσης θα ήθελα να ξέρω πόσος χρόνος χρειάζεται για τις ε, αδειοδοτήσεις που δίνονται σε σιδηροδρόμους αυτή τη στιγμή από πλευράς του οργανισμού. Προς το παρόν, ε, λόγω προστατευτισμού φτάνουμε σε 18-23 μήνες, πραγματικά σκανδαλώδεις ημερομηνίε. Ε, πόσο καθυστερεί αυτή τη στιγμή ο οργανισμός. Και τέλος, υπάρχει ένα πρόβλημα και στην Ισπανία ε, για τα, τις προστατευτικές δικλείδες στα τρένα, τα οι οποία δεν βρίσκονται στο ύψος της νομοθεσίας και ο κόσμος πεθαίνει λόγω της έλλειψης προστασίας. Ξέρω ότι υπήρξαν προειδοποίησεις προς την Ισπανία. Θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς θεωρείτε ότι προχωρούν στην επίλυση αυτού του τεράστιου προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου. Η κυρία Λεσόντε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, στην, ε, στα πρόθυρα της έναρξης ανταγωνισμού των υπηρεσιών ε, στους σιδηροδρόμους στη Γαλλία θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται με το άνοιγμα σε χώρες οι οποίες ήδη έχουν προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Ε, εμπορικές υπηρεσίες, ε, υπηρεσίες προώθησης που σημαίνει ότι υπάρχει ε, ε, μεγάλη εδαφική και κοινωνική σημασία την οποία δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε. Δεν είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία, ιδίω αν λάβουμε υπόψη και το επίπεδο ασφαλεία, το κόστο εκμετάλλευση ανά χιλιόμετρο, καθώ επίση και την αύξηση των ε, εισιτηρίων. Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 Αραφέρ, ε, υπάρχει ενδιαφέρον των ε, επενδυτών ε, μεταξύ των συμβατικών και των ε, μη συμβατικών τομέων. Όσον αφορά τις εσωτερικές υπηρεσίες, μόνο έξι χώρες άνοιξαν τον ανταγωνισμό, αλλά στην πράξη γίνεται μόνο για τις μη συμβατικές υπηρεσίες. Επομένως, θα πρέπει ο οργανισμό σιδηροδρόμων να ελέγξει αυστηρά το άνοιγμα του ανταγωνισμού του τομέα των σιδηροδρόμων και επίση να ελέγξει και του κοινωνικού εταίρου και του εκπροσώπου των ταξιδιωτών, διότι δεν θα πρήκεται να γίνε θα γίνονται αυτά ει βάρο των εργαζομένων. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πάρα πολλέ ερωτήσει. Διάρκεσε πολύ η διαδικασία των ερωτήσεων θα ήθελα και εγώ να σταθώ στην, ε, στον τομέα της ασφάλειας. Είναι πραγματικά η προτεραιότητα της Επιτροπής μας. Ξέρετε ότι η ασφάλεια είναι ε, σκέλος και των δικών σας των ευθυμών και δεσμεύσεων και υπάρχει και ένα θέμα το οποίο δεν συζητήθηκε παρά το γεγονός ότι αναφέρομαστε σε άνοιγμα του ανταγωνισμού και ορισμένες φορές υπάρχουν και κοινωνικές συνέπειες οι οποίες πρέπει να λάβουμε υπάψη. Υπάρχουν και άλλε χώρε οι οποίε ε, δεν ενδιαφέρονται καθόλου με τις, για τι κοινωνικέ συνέπειε ε, ε, στις δημόσιες συμβάσεις, για παράδειγμα, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους μισθούς, να υπάρχουν κατάλληλες αποζημιώσεις κλπ. Το θέμα είναι όμως πώς θα μπορέσετε κι εσείς να προλάβετε τις ε, διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των επιβατών. Όταν λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν, για παράδειγμα, 8 ποδήλατα σε κάθε τρένο. Ε, αυτά θα είναι ουσιαστικά ερωτήματα και όπως είπε και ο κύριος ε, Ρικέ, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τον έλεγχο του προσωπικού, διότι αναφέρθηκε και το υπενθυμίσαμε, αν δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα, δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ποδήλατα στα τρένα, δεν θα έχουμε ε, συνδυασμένες μεταφορές και δεν προχωράμε τη διαλειτουργικότητα. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ήθελα να μου απαντήσετε και σε αυτό το ερώτημα. Πρέπει να προλάβουμε και κάπως τα πράγματα. Έχετε το λόγο κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους ε, για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το τέλος. Θα απαντήσω πρώτα στην ερώτηση για τις ιδιωτικοποίησεις. Καταρχάς πρέπει να δηλώσω ότι οι οικονομικές πτυχές δεν είναι ε, στην εντολή του οργανισμού. Εάν εξετάσουμε μόνο τους τομείς ε, στους οποίους παρακολουθούμε εμείς την κατάσταση, που είναι η ασφάλεια των σιδηροδρόμων, δεν βλέπουμε κάποιο αρνητικό στοιχείο για το κατά πόσον ε, η υπηρεσία είναι ιδιωτική ή δημόσια. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να μιλήσω για τις πιο γενικές πτυχές που αναφέρατε. Όσον αφορά την ασφάλεια όμως, ε, φαίνεται ότι υπάρχει και κάποιος θετικός αντίκτυπος από την ιδιωτικοποίηση, αλλά αυτό βέβαια είναι ακόμα προσυζήτηση. Όσον αφορά τις ερωτήσεις της κυρίας Μπιλμπάου. Καταρχάς, γιατί ο χρόνο διοδότησης. Υπάρχουν αυστηροί νομικοί περιορισμοί στην οδηγία της ε, διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων και τη διαδικασία της αδειοδότησης. Για να δοθεί λοιπόν νέα άδεια, έχουμε 8 μήνες για να δηλώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος και από εκεί και πέρα έχουμε 4 μήνες για να λάβουμε απόφαση. Είτε θετική με έγκριση της άδειας ή αρνητική απόφαση και απορρίπτεται η αίτηση. Ε, υπάρχει λοιπόν αυστηρός περιορισμός όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Για τους πρώτους δυόμισι μήνες ε, που ε, ε, δόθηκαν 92 άδειες, στην πραγματικότητα πρόκειται για έγκριση τύπου. Και σε αυτή την περίπτωση της έγκρισης τύπου υπάρχει ένα νομικό όριο ενός μηνός αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο έχουμε κάτι λιγότερο των 15 ημερών. Είμαστε στο ίμιση λοιπόν του νομικού ωραίου και η φιλοδοξία είναι του χρόνου τουλάχιστον να είμαστε στις 7 ημέρες. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας όσον αφορά το χρόνο έγκρισης. Για την ερώτησή σας τώρα για το κατά πόσο είμαστε αισιόδοξοι ε, αν τα κράτη-μέλη θα μεταφέρουν τη νέα δέσμη μέτρων, ένας από τους λόγους στην Ισπανία ήταν η πολιτική κατάσταση στην Ισπανία, όχι οι συγκεκριμένε σιδηρόδρομοι. Ε, είχαμε εκλογέ, νέα κυβέρνηση κλπ. Αλλά είμαι αισιόδοξο ε, και πιστεύω ότι η μεταφορά θα γίνει το 2020. Αντιστοίχω για χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο ή την Αυστρία, την Πολωνία, πιστεύω ότι οι χώρε αυτέ είναι όλε σε καλό δρόμο και θα ε, δούμε τις χώρες στο σύστημα του χρόνου. Ετέθη μια ερώτηση για το κατά πόσον κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα ανοίγματο ε, τροχών για τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. Εδώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο, διότι υπάρχει το ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά είναι το 1435 που είναι συνήθι, το σύνηθες άνοιγμα, αλλά υπάρχει και ένα ε, σύστημα το 1520 στην ερώτηση του κυρίου Γιούρες απαντώ, το οποίο ε, το ελέγχει η Ρωσία και θα υπάρχει πάντα αυτό το 1520 και το ερώτημα είναι μέχρι ποιο σημείο θα διεισδύσει στην Ευρώπη αυτό το 15-20 και μέχρι ποιο σημείο θα είναι εκτός Ευρώπης. Υπάρχει και μία ερώτηση όσον αφορά τη μείωση των εθνικών κανόνων και ε, θα μπορούσα να έχω και συγκεκριμένα στοιχεία, τα είχα ετοιμάσει σε μια διαφάνεια, δεν τα είχα. Δυστυχώ. μπορώ να σας δώσω προφορικά τα στοιχεία. Ξεκίνησε μια πρωτοβουλία πολύ αυστηρών κανόνων, μείωσή τους το 2016 και τότε είχαμε 14.312 κανόνες, όχι 11.000 αλλά 14.312 κανόνες. Ε, εθνικούς κανόνες για έγκριση οχημάτων. Μόλις ολοκληρώθηκε μία έκθεση για τη μείωση αυτών των κανόνων ε, το 2019 και τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι 1026. Μειώσαμε δηλαδή από πάνω από 14.000 στους 1.000. 300-400 είναι ακόμα σε συζήτηση και Ο οργανισμό δεν συμφωνεί με τα κράτη-μέλη ότι είναι απαραίτητοι αυτοί οι κανόνε. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα να φτάσουμε στον αριθμό που αναφέρατε εσεί, μερικέ εκατοντάδε. Ε, εθνικούς κανόνες. Αλλά πιστεύω πραγματικά ότι το γεγονός ότι πήγαμε τους 14.000 στους 1.000 είναι πραγματικά πολύ μεγάλο επίτευγμα. Για να σας δώσω μια εικόνα, στο TSI, που είναι η Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή, έχουμε ακριβώς 531 κανόνες. Το κράτος μέλος που έχει τον υψηλότερο αριθμό ε, εθνικών κανόνων είναι η Ιταλία που έχει λιγότερους από 100. Έχουμε λοιπόν 500 ευρωπαϊκούς κανόνες και 100 εθνικού κανόνες τώρα. Πριν είχαμε χίλιους και εθνικούς κανόνες και μόνο 531 ευρωπαϊκούς κανόνες. Έχουμε αναστρέψει εντελώ την κατάσταση λοιπόν. Τώρα, για να απαντήσω στην κυρία Τάλερ για το κόστος. μπορούμε να εκτιμήσουμε σαφώς το κόστος αυτών των διακοπών στα σύνορα ε, για τη λειτουργία. Και υπάρχει μια παρέμετρο. Είναι πρώτον θέμα χρόνου. Διότι αν κάποιο χάσει τρει ώρες ή την Παρασκευή μπορεί να χάσει και 48 ώρες, τότε πρόκειται για τεράστια οικονομική απώλεια. Και αυτό το οποίο είναι ακόμα πιο ενοχλητικό είναι το γεγονό ότι δεν υπάρχει προβλεψιμότητα. Διότι αν στέλνει ένα εμπόρευμα με ένα φορτηγό, ξέρει ε, με ακρίβεια 15 λεπτών πότε φτάνει το εμπόρευμά σου. Με το τρένο δεν το ξέρει ούτε καν εντό 24 ερών. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όσον αφορά το κόστο. Το κόστος μόνο για το σύστημα σηματοδότησης, το οποίο είναι διαφορετικό σε κάθε χώρα, είναι πάρα πολύ ψηλό. Αν δείτε το Eurostar που πηγαίνει από το Λονδίνο στο Παρίσι και στο Άμστερνταμ. Αυτό το τρένο το Eurostar έχει 9 διαφορετικά συστήματα σηματοδότησης να περάσει. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 9 συστήματα είναι 9 φορές πιο ακριβά από ένα σύστημα. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε μια εκτίμηση του κόστους. Τώρα, για να απαντήσω στον κύριο Ρικέ Πρώτα, για τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη σιδηροδρομική σύνδεση Βαλενσιέν-Βρυξέλλες. Αυτή τη στιγμή όλες οι συνεδριάσεις ε, με τις ε, ομάδες εργασίας γίνονται στη, ΛΥΛ. στη και συνήθως έχουμε 25 με 50 άτομα στη συνεδριάσεις κατά μέσο όρο και έχουμε όλο ένα και περισσότερους ετούντες που έρχονται στη Βαλενσιέν για να συζητήσουν ε, την υποψηφιότητά τους. Νομίζω λοιπόν ότι το λογικό ε, στοιχείο είναι ότι θα υπάρχει ε, χρήση ε, της γραμμής Βαλενσιάν-Βρυξέλλες. Τώρα, όσον αφορά τις προσλήψεις, με τον νέο κανονισμό και στον τεχνικό πυλώνα έχουμε λύσει το θέμα των μόνο προσωρινών συμβάσεων. Μπορούμε πλέον να παρέχουμε μόνιμη σύμβαση, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και εν μέρη ήμασταν πολύ τυχεροί τους τελευταίους ε, μήνες γιατί μπορέσαμε να προσελκύσουμε ε, πολύ καλούς ανθρώπους ε, από τον κλάδο που εργάζονται πλέον για μας. Έχουμε κάποια προβλήματα ακόμα να προσελκύσουμε άτομα με τις σωστές γλωσσικές δεξιότητες. Δεν έχουμε, για παράδειγμα, γερμανόφωνους εμπειρογνώμονες και πολωνούς εμπειρογνώμονες. Έχουμε γαλλόφωνους, Ιταλούς, Ισπανούς, δεν είναι πρόβλημα αυτό, αλλά μας λείπουν κάποιες άλλες ε, γλώσσες. Ο κύριος Πίπερ ρώτησε για τη μεταφορά. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα ποιότητας της μεταφοράς της οδηγίας. Νομίζω ότι θα το δούμε του χρόνου όταν θα έχουμε και τις νέες χώρες, τις υπόλοιπες χώρες και από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τις παραβάσεις. Ο κύριος Ζήλε ανέφερα ήδη τη μείωση των κανόνων. Πλέον από 14.300 είμαστε στους 1.000 και ε, το 15-20 άνοιγμα τροχών, νομικός ναι και ε, τα βαγόνια του 15-20 με άνοιγμα 15-20 πρέπει να ε, έρχονται σε εμά. αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δώσει αδειοδότηση για βαγόνια 15-20 συζητούμε τις τέσσερις χώρες, ε, τις τρεις Βαλτικές και τη Φιλανδία. Η Φιλανδία είναι μία από τις ε, χώρες που βρίσκονται στο πρώτο σκέλος. Ε, υπογράψαμε συμφωνία συνεργασίας με τη Φιλανδία. Είμαστε σε συζητήσεις σε καλό στάδιο με τις χώρες της Βαλτικής και πρέπει εκεί όχι μόνο να συνάψουμε ε, ατομικές ε, συμβάσεις συνεργασίας, αλλά και μια συνολική σύμβαση συνεργασίας, ειδικά για το 15-20. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι μόλις ανανεώθηκε η Συμφωνία Συνεργασίας με τον αρμόδιο οργανισμό των χωρών ε, με άνοιγμα τροχών 15-20 και έχουμε και τακτικές ανταλλαγές απόψεων και με αυτούς. Τώρα, για την ερώτηση για την Ιταλία. Έχουμε δύο πτυχές εδώ. για τις διασυνοριακές μεταφορές. Το ένα είναι η αδειοδότηση των τρένων και εδώ έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό με τους συναδέλφους από τον κλάδο και υπάρχει και το θέμα του πιστοποιητικού ασφαλείας. Η Τρέν Ιτάλια μας προσέγγισε για ένα πιστοποιητικό ασφαλείας το οποίο θα επιτρέπει τη μεταφορά ε, διασυνοριακά. Μετά, το ερώτημα για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ετέθη αρκετές φορές, αν δεν κάνω λάθος. Απάντησα προηγουμένως. Για την Ισπανία τώρα, πρώτα, πρώτα, είχαμε άμεση εμπλοκή με τις Ισπανικές αρχές, με τη Ρέμφε κυρίως και την Άντιφ, ε, έγινε μια εις βάθος ε, διαδικασία ελέγχου πέρσι με την Ισπανία για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με το επίπεδο συνεργασίας ε, και το ανοιχτό πνεύμα. Θεωρώ ότι ένα πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Αρχής είναι ότι εμείς είμαστε ουδέτεροι, είμαστε ανεξάρτητοι, δεν έχουμε πολιτική ατζέντα σε καμία χώρα και μπορούμε απλώς να βασιστούμε σε απτά στοιχεία και πρέπει να πω ότι η συνεργασία, το ανοιχτό πνεύμα, η εμπιστοσύνη, διότι ούτως ή άλλως η ασφάλεια είναι πάντα θέμα εμπιστοσύνης, έχει βελτιωθεί και είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Κατόπιν, ο κύριος Μαρινέσκου με ρώτησε για την ενιαία θηρίδα. Αυτή τη στιγμή εκτός από τα εμπορικού εμπορικούς σειρμούς, γιατί για τα εμπορικά δεν περιορίζονται σε ένα διάδρομο, γινόμαστε, γίνονται για όλη την Ευρώπη. Η άλλη μεγάλη κατηγορία σειρμών που έχουμε είναι ε, είναι οι μηχανέ και εκεί έχουμε μόνο τι κάτω χώρες, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Δεν μπορούμε πραγματικά να δούμε ποιοι θα είναι οι διάδρομοι, θα τους δούμε το 2020 όταν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ε, θα ενταχθούν στο σύστημα. Η δεύτερη ερώτησή σας είναι αν υπάρχει ένα πλήρες σχέδιο για τη μείωση των εθνικών κανόνων. Η απάντηση είναι ναι. Σας έδωσα το παράδειγμα της μείωσης ε, των κανόνων για την έγκριση των οχημάτων που ήταν η πιο επίγουσα ανάγκη διότι έπρεπε να ξεκαθαριστεί το σύστημα ε, πριν προχωρήσει η διαδικασία και ταυτόχρονα προχωράμε και τους κανόνες ασφαλείας. Εκεί έχει επιτευχθεί ιδιαίτερη πρόοδος και προχωρούμε επίσης και τους κανόνες για τη λειτουργία. Οι κανόνες λειτουργίας είναι ίσως πιο δύσκολο θέμα διότι εδώ υπάρχουν και προβλήματα όπως για παράδειγμα η επιχειρησιακή γλώσσα. Ε, αμέσως λοιπόν τίθενται και κάποια πολιτιστικά ζητήματα. Ε, έχουμε σχέδιο, συνεχίζονται οι εργασίες, αλλά για να ενερμανιστούν πλήρως ε, τα θέματα λειτουργίας έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά. Ελπίζω να κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Ε, αν όχι, παρακαλώ, ελεύθερο επενθυμίστε μου. Ευχαριστώ πολύ τον Διευθυντή του οργανισμού, τον κύριο Ντόπελμπάουερ. Πραγματικά μας παρουσιάσατε όλα τα θέματα. Επιστήσατε και την ε, προσοχή μας σε αυτά που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό για τον οργανισμό σας. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, πρέπει να βλέπουμε μακριά, να έχουμε όραμα. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω να επεξεργαστώ μαζί με την Επιτροπή ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανανέωσης και ανακαίνησης των ε, σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Είμαστε σε θέση με το Invest Europe να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το χρειάζονται όλοι και είναι κάτι που είναι χρήσιμο και επωφελές και για το κλίμα και για την βιομηχανία αλλά και στη δική μου περιοχή, κοντά μάλιστα και στην περιοχή του κυρίου Ρικέ, ο οργανισμός σας, θα έρθουμε και θα σας δούμε και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει άμεση σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ μαζί μας, αγαπητοί συνάδελφοι. Ολοκληρώσαμε τη συνεδρίασή μας και θα σας βρω αύριο στις 9 οι συντονιστές. Μην ξεχάσετε, οι ψηφοφορίες αρχίζουν στις 10. Μην ξεχάσετε και τις κάρτες σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Διευθυντή του Ήρα. Τον χειροκροτούμε.